Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη της συνεδρίασής μας. Εγκρίνεται η μέρη σε διάταξη αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και τα πρακτικά της 29ης Αυγούστου θα θεωρηθούν εγκεκριμένα αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις και να αρχίσουμε με το πρώτο κυρίως θέμα της τη διάταξης, την έκθεση πρωτοβουλίας ό,τι αφορά το σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα. Έκθεση πρωτοβουλίας και σχέδιο γνωμοδότησης προς την Επιτροπή ΕΦΕΤ. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή μας, το συντάκτη γνωμοδότησης μάλλον, και μετά στους κοιόδης εισηγητές. Και θα ήθελα και τη γνώμη μετά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Τελίσκα, πολύ καλημέρα σας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Δεν θα ήθελα να επαναλαμβάνομαι. Ε, είναι σύντομες όλες οι γνωμοδοτήσεις, το ξέρετε, δεν θα διαβάσω το περιεχόμενό της. Το θέμα είναι απλό για πολλούς από εμά, αλλά για κάποιους ίσως είναι λίγο προβληματικό ή για κάποιες πολιτικές ομάδες ίσως. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Ε, παρόλο που η έκθεση αναφέρεται στην στρατιωτική κινητικότητα, αναφέρεται σε διπλή χρήση, πολιτική και στρατιωτική. Αυτό σημαίνει, επειδή έχουμε και στρατιωτική κινητικότητα, αν σε φάση σχεδιασμού ε, και στη συνέχεια, στην κατασκευή ή στην προσθήκη προστιθέμενης αξίας σε υπάρχουσα υποδομή, αυτό γίνεται για λόγους ε, ε, στρατιωτικούς. Αυτό το νόημα έχει το στρατιωτικό. Αλλά όλοι είμαστε εξαρτημένοι από τις στρατιωτικές μας ικανότητες που αν παραστεί ανάγκη, είτε για προληπτικούς λόγους είτε για αμυντικούς, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να μετακινήσουμε βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι οι υποδομές αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά ανάγκη και αμυγός για στρατιωτικούς σκοπούς. Θα μπορούσαν κάλλιστα να εξυπηρετούν οι υποδομές αυτές ε, και πολιτικούς και στρατιωτικούς σκοπούς σε περιπτώσεις ε, κατεπίγουσας ανάγκης, για παράδειγμα, εκεί που πρέπει να μετακινήσουμε μεγάλο τμήμα εξοπλισμού ή σημαντικά στοιχεία πολύ γρήγορα μας εξυπηρετούν τέτοιες υποδομές και σε αυτό το σημείο δίνουμε έμφαση στο σχέδιο γνωμοδότησης. Μιλάμε κυρίως για διπλή χρήση, πολιτική και στρατιωτική. Αυτό που λέω ξεκάθαρα στο σχέδιο γνωμοδότησης είναι ότι επουδενή δεν θα επικεντρωθούμε μόνο σε αμυγός στρατιωτικά σχέδια και προγράμματα. Θέλουμε να λάβουμε υπόψη και άλλους πιθανούς ε, σκοπούς μεταφοράς επιμελητίας, ε, μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η επιβατων και ουτω αυτη ειναι η λογικη της έκθεσης, ο διπλός σκοπός, διτή χρήση. Επίσης, θέλουμε να αποφύγουμε ε, για αμυγό στρατιωτικούς λόγους να χρειαστεί να τροποποιηθεί οποιοδήποτε σχέδιο σε οποιαδήποτε φάση του, γιατί κάτι τέτοιο θα αυξήσει το κόστος. Οπότε θα πρέπει σε συγκεκριμένες φάσεις όταν μιλούμε για το σχέδιο δράσης να υπογραμμίσουμε ότι από τα πρώτα στάδια, από τα πρώιμα στάδια να έχουμε σημαντική ενιολογική προσέγγιση. Νομίζω ότι είναι πολύ θετική η γνωμοδότησή μας. Ευθυγραμμίζεται και με τις πολιτικές μας αποφάσεις και η κρατούσα θέση είναι ότι Πρόκειται για σημαντική ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα κόσμο που γεωπολιτικά γίνεται όλο και πιο περίπλοκος. Δεν χρειάζεται να σας πω τις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι όλοι έχουμε επίγνωση αυτού του θέματος. Αυτά λοιπόν είναι τα εισαγωγικά μου σχόλια, κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που σας αναπτύσσω το θέμα αυτό και στα πλαίσια του συνδέοντας στην Ευρώπη. Ε, είχαμε σταθεί και στο ζήτημα αυτό. Θα ήθελα πάντως να πω ότι το κονδύλιο για τα στρατιωτικά θέματα δεν είναι ένα παράρτημα ή ένα τμήμα που διαχωρίζουμε από το συνδέοντα στην Ευρώπη. Ουσιαστικά συμπεριλαμβάνουμε στο συνδέοντα στην Ευρώπη συμπληρωματικούς πόρους για τα στρατιωτικά θέματα. Και οι βασικές αρχές και διατάξεις για το συνδέοντα στην Ευρώπη ελπίζω να διαθετηθούν όσον ούπο και να εφαρμοστούν αμέσως και στο στρατιωτικό σκέλος που επαναλαμβάνω είναι προσθήκη με επιπλέον κονδύλια. Αυτά και είμαι στη διάθεσή για τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε κύριε Τελίτσκα. Μήπως θα μπορούσατε να μας υπενθυμίσετε τα ποσά. Είναι 6-6,5 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Παρα... Παρακαλώ δεν άκουσα. Ποιο είναι το κονδύλιο αυτής της δημοσιονομικής γραμμή. 6 ή 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. ...6,45 δις. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ο κύριος Βαντεκάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον συνάδελφο Μαρινέσκο, που είναι αρμόδιος για το θέμα αυτό και βρίσκεται στη Βιέννη αυτή τη στιγμή, στην ε, συνεδρίαση του Προεδρείου του ΕΛΚ. Εκείνο στη Βιέννη και εγώ εδώ. Βλέπετε πόσο με έχει καταβάλει αυτό το γεγονός. Διαβάζετε τη θλίψη στο πρόσωπό μου. Ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφο Τελίτσκα, λέει ο κύριος Μαρινέσκου, Ευχαριστεί τον κύριο Τελίσκα για την γνωμοδότησή του και τον ενημερώνει ότι σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε με τη στρατηγική του κύριου Τελίσκα. Ο Πάβελ και ο Μάριαν είναι συνεισηγητές. Ε, κάτι που διευκολύνει τα πράγματα για ένα άλλο θέμα πότε συμβάλλει στην εξορόψη του κειμένου. Πάβελ, στάθηκες στο ζήτημα της διτής χρήσης, πολιτικής και στρατιωτικής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και έχω μία ερώτηση εδώ, μία απορία. Εγώ ε, εκείνο από την αφετηρία ότι όταν μιλούμε για διτή χρήση υπερέχει το πολιτικό σκέλος, το μη στρατιωτικό και η πολιτική μη στρατιωτική χρήση και οι αντίστοιχοι λόγοι και στόχοι. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η δίτη χρήση. Μιλάμε για έναν προϋπολογισμό 6,45 δισεκατομμύρια. 6,5 έλεγε η αρχική πρόταση και ελπίζω να διαφυλάξουμε αυτό το προϋπολογισμό. Και μάλιστα, αν κατάλαβα καλά, πριν τις 31 Δεκεμβρίου του 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τα σχέδια αυτά. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως είναι κάπως περίεργο που μιλάμε τόσο εύκολα για στρατιωτικούς ε, στόχους, σκοπούς. Θα προτιμούσα να μιλούμε περισσότερο για ειρηνευτικούς σκοπούς. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ευχαριστώ πάντως τον Πάβελ, τον Μαριάν Μαρινέσκου και παραλαμβάνω ότι σε μεγάλο βαθμό το ΕΛΚ συμφωνεί με την γνωμοδότηση. Θα δούμε βέβαια στην πορεία τι τρόποι θα πάρουν διαπραγματεύσει. Ευχαριστούμε. Κύριε Βαντενκάμπ. Κυρία Γκραπίνη έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την Επιτροπή που με βοήθησε στο έργο μου σκιώδους συγκεκριές. μου έδωσε τη δυνατότητα της επικοινωνίας ε, ως προς το σχέδιο δράσης για την ε, πρόταση. Ευχαριστώ τον ε, συνάδελφο κύριο Τιλίτσκα επίσης για το σχέδιο γνωμοδότησης αλλά και για τις εξηγήσεις που μας έδωσε. κάναμε μια ομάδα εργασία. Ε, ρωτούσε ο κύριο Φαντεν Κάμπ νωρίτερα γιατί στρατιωτική, γιατί αναφορά στη στρατιωτική χρήση. Πρέπει να το σκεφτούμε βεβαίω καλά, αλλά. Υπάρχει, βέβαια, ίσως όταν κάτι δεν μας αρέσει δεν θέλουμε και να το συζητούμε, αλλά εάν υπάρχει δεν πρέπει να το αναφέρουμε. Και στα όσα είπαν οι κύριοι Τρίτσκα και Φαντεν Κάμπ έχουμε αυτή τη λέξη κλειδί, διπλή χρήση, διτή χρήση. Ε, έτσι λοιπόν αυτό το υλικό δεν έχει μόνο στόχο την εξυπηρέτηση πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Ε, γιατί πολύ συχνά ε, ομάδες ε, στρατιωτικών με υλικό στρατιωτικό κινητοποιούνται για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση φυσικών κρίσεων. Και εδώ περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται για ενσωμάτωση σε πολιτικές χρήσεις των στρατιωτικών ε, δυνατοτήτων. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στους ε, πολίτες. Είναι δυνατόν να πούμε ότι χτίζουμε μία γέφυρα που θα χρησιμοποιεί μόνο ο στρατός και μία που θα χρησιμοποιούν μόνο οι πολίτες ή ένα δρόμο που θα χρησιμοποιεί μόνο ο στρατός και μόνο οι πολίτες. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτή την ε, ενσωμάτωση λοιπόν των μέσων και των έργων για να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα και σε οικονομικούς όρους και να ενισχύσουμε την ασφάλεια των πολιτών. Μην φοβόμαστε τη λέξη ασφάλεια. Έχουμε καθήκον να ε, προασπιζόμαστε και να ενισχύουμε την ασφάλεια των πολιτών. 6,5 όχι 6,35 κύριε Τελίτσκα, είναι το ποσό που έχω εγώ υπόψη. Αλλά τελικά δεν είναι αυτό που μετράει. Μετράει το πώς θα δαπανηθούν τα κονδύλια αυτά. Πώς θα ενσωματωθούν στα ε, διευρωπαϊκά δίκτυα, ε, στους ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρες, χωρίς βέβαια να επηρεάσουν αρνητικά τις εμπορικές μεταφορές. Και έχω κάνει λόγο για την περιγραφή των μεταφορών εμπορευμάτων, επικίνδυνων εμπορευμάτων λοιπά, Η στρατιωτική χρήση που οπωσδήποτε θα πρέπει να μεταφέρονται κάποια στιγμή. Και προβλέπεται κάτι σχετικό. Βέβαια κάποιοι θεωρούν ότι η έκθεση είναι τεχνική, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι πολιτικού χαρακτήρα περισσότερο νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Με τον εισηγητή, με τους συναδέλφους και της δικής μου της ομάδας, ακόμη για να διατυπώσουμε τροπολογίες που θα μας επιτρέψουν να περιγράψουμε τα ζητήματα και να εξασφαλίσουμε την ε, συμπερίληψη στο σχεδιασμό μας και τη στρατιωτικής κινητικότητας. Δεν μπορούμε να την παραγνωρίσουμε, δεν μπορούμε να την βάλουμε στο περιθώριο, όπως και την πολιτική κινητικότητα την χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ κύριο και έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι γενικώ στηρίζουμε την πρωτοβουλία αυτή για την εθέτηση ε, κάποιων υποδομών μεταφορών για τη στρατιωτική κινητικότητα. Και όντως, αν θέλουμε ειρήνη, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για πόλεμο. Και ιδιαίτερα όταν έχουμε εμπόλεμε συγκρούσει στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προσαρμογή των ε, διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών ε, για στρατιωτικού σκοπού. Μέχρι στιγμή ε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών ε, είχαν αποκλειστικά πολιτική χρήση. Και οπότε θα πρέπει να κάνουμε νέο ε, προγραμματισμό και θα πρέπει σε μόνο έκτακτες περιπτώσει. να υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης χρηματοδότηση υποδομών μεταφορών που δεν περιλαμβάνονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και για αυτού του σκοπού. Έτσι θα διευκολύνουμε τη στρατιωτική κινητικότητα και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε λίγες παρατηρήσεις για τους τρόπους χρηματοδότησης. Να δούμε πώς θα κατανοίγουμε τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων σχεδίων και ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής των ε, σχεδίων. Ε, στα πλαίσια του Συνδέοντα στην Ευρώπη έχουμε διαδικασία ανταγωνισμού, με υποβολή προσφορών και διαγωνισμό. Θα πρέπει να δούμε ε, μήπως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχουν ε, οι προμήθειες στρατιωτικές ε, μεταφορές. Επίσης, ε, 30% να έχουμε για τα επενδυτικά σχέδια, 50% για τα διαρθρωτικά, να έχουμε ένα ποσοστό για τα διασυνοριακά σχέδια, να δούμε υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις θα εγκρίνονται αυτά τα σχέδια, το επίπεδο συμπληρωματικής χρηματοδότηση ε, του Συνδέοντος τη Ευρώπη ε, ίσω ε, δεν ανταποκρίνεται στου ιδιαίτερου στόχου που έχει ένα σχέδιο στρατιωτική κινητικότητα. Όλε αυτέ οι ιδιαιτερότητες θα πρέπει να, τα, να τις λάβουμε υπόψη και κύριος ο συντάκτης γνωμοδότης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σλοτόσκι. Κύριε Γιάνντε, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προτιμούσαμε το θέμα της στρατιωτικής κινητικότητας να μην ήταν μέρος του ΣΕΦ. Είναι σημαντικές και οι ανάγκες της πολιτικής προστασίας. Και έχουμε ε, για τα 645 εκατομμύρια που θα φύγουν από το ΣΕΦ. Θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών πάνω απ' όλα. Αλλά δεν είναι και σαφές ακόμη πώ θα εκτελεστούν τα κονδύλια αυτά. Δεν έχουν αναλυθεί αρκετά τα έργα που ε, έχουν προτείνει τα Υπουργεία Άμυνα. Νομίζουμε ότι πρώτα πρέπει να επιληθεί το θέμα της διασυνοριακή συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των στρατιωτικών υποδομών. Όμω δεν υπάρχει αρκετή έμφαση στην δυτή χρήση και τα κριτήρια αντιστατοτική κινητικότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Νταλούντα. Κύριε Βαντάρλεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην παράγραφο 2 του σχεδίου γνωμοδότησης, ο εισηγητής τοποθετείται ξεκάθαρα υπέρ του σχεδίου. Εγώ όμως έχω κάποιες επιφυλάξεις, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι σε, κάποιες, ε, σε κάποια σημεία του κειμένου δεν είναι αποτελεσματική διατύπωση. Όταν μιλάμε για τη διτή χρήση, πρέπει να βρούμε τη σωστή, το σωστό συσχετισμό μεταξύ της θεωρητικής και της πολιτικής συνιστώσας. Στα αεροδρόμια έχουμε διτή χρήση πολλές φορές. Υπάρχει μια συνιστόσα στρατιωτική σε κάποια αεροδρόμια που είναι και πολύ ε, παρούσα, πολύ έντονη παρουσία της και αυτό βαρύνει στη ζυγαριά. Μιλάμε για υποδομές όμως που είναι κατά κύριο λόγο πολιτικού χαρακτήρα ε, και θα πρέπει να δούμε αν μπορούν να έχουν χρήση στη δοχή. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα κατανεμηθούν και τα έργα. Τα έργα που αποσκοπούν ε, στην δυτή χρήση και μόνο και έχουν και συγκεκριμένο κόστο. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώ θα τα διαχειριστούμε τα έργα αυτά. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά που ε, σκοπό έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα του κλίματο, του περιβάλλοντο ή την μεταφορά εμπορευμάτων. Εκεί θα ήθελα λίγο περισσότερε εξηγήσει. Και τρίτη παρατήρηση, κάτι πολύ σημαντικό επίση και κανεί δεν το σχολίασε ω τώρα. να δούμε τι γίνεται με την ε, πρωτότυπη αυτή νομοθεσία, αυτό που λέμε την ε, καμπούρα της καμήλας, όπως λέμε σε κάποιες γλώσσες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, προφανώς και μια καινούργια, ε, ένα καινούργιο νομοθέτημα εκπλήσει, αλλά εκπλήσει με τα προφανή. Θα πρέπει να κοιτάξουμε με την νομοθεσία που προτείνουμε, να μην κατατεμαχίσουμε τον επιδιωκόμενο στόχο. Με μια φέτα σε ένα νομοθέτημα από εδώ, μια άλλη φέτα του σαλαμιού σε ένα νομοθέτημα από εκεί και ούτω καθεξής. Κυρία Πρόεδρε, λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε μια πιο κριτική στάση στην όλη εξέταση του σχεδίου. Ευχαριστούμε κύριε Φαντάλεν. Κυρία Ντεμόντα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ τον εισηγητή για την πρότασή του. Πρέπει βέβαια να θεωρήσουμε σημείο αφετηρία στην ανακοίνωση της Επιτροπής και το σχέδιο έκθεσης της ΑΦΕΤ, όπου νομίζω βλέπουμε κάποιες σαφείς κατευθύνσεις. Η διτή χρήση βέβαια αναφέρεται, αλλά τελικά γίνεται ρητή αναφορά στην στρατιωτική χρήση. Έτσι λοιπόν δεν νομίζω ότι μπορούμε να ε, εξαντλήσουμε το επιχείρημα στο ότι πρόκειται για τεχνικούς όρους και τεχνική τοποθέτηση. Έχουμε να κάνουμε με ζητήματα βαρύνοντα πολιτικά και κυρίως το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι αυτοί, τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σε τι έργα. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μπορούν να εκτιμηθούν με προσοχή ως προς το στόχο τους και αναφέρθηκε νωρίτερα και η στόχευση, οι γέφυρες δηλαδή και οι παραμεθόριες περιοχές. Βεβαίω έχουμε θέμα και με το χρονοδιάγραμμα, καθώς το 18 ήδη τρέχει και έχουμε μόλις το έτος 2019 ακόμη για να ολοκληρώσουμε το σχεδιασμό αυτό και νομίζω ότι θα έπρεπε να μιλήσουμε γενικότερα για ενίσχυση υποδομών έτσι ώστε να βάλουμε και μια σουρντίνα στις λοιπές ε, ε, επιλογές. Γιατί όταν μιλούμε για αποτροπή ή αποτρεπτική χρήση, αμέσως δίνουμε την εικόνα ότι η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει επιθέσεις. Επίσης, χερσαίες επιθέσεις νομίζω δεν είναι δυνατόν να συζητούνται στην ε, εποχή που ζούμε δεν είναι τόσο επίκαιρη δηλαδή η άμυνα μέσω, με, με στρατόξυρας. Ε, επίσης ήθελα να δούμε και με τον εισηγητή τι εννοεί ως παραμεθόριες περιοχές. Μιλούμε παραμεθόριο μεταξύ δύο κρατών μελών ή παραμεθόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ε, Ανατολική Ευρώπη, παραδείγμα τις χώρε ε, που βρίσκονται στα ανατολικά της Ευρώπης. Ε, θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις από τον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ, πολύ σύντομα. Έχεις δίκιο ότι την ειρήνη την εξασφαλίζουμε μόνο όταν είμαστε έτοιμοι και για την άμυνα. Ναι. Γιατί όμως πρέπει ο τομέας των μεταφορών να δώσει 6 δισεκατομμύρια για υποδομές στρατιωτικές. Όταν λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για υποδομές, τότε αυτά θα πρέπει να αναπτυχθούν, να αντληθούν σε πεδογενικό και να διατεθούν σε πεδογενικό. Δεν μπορούμε να λέμε ότι μόνο οι, οι μεταφορές δίνουν ένα τέτοιο ποσό 6 δισεκατομμύρια μόνο για στρατιωτική χρήση. Στη τελευταία ανάλυση θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει ε, το Ταμείο Γιουνκέρ να δώσει το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, όχι να δοθεί εντύπωση ότι εμείς έχουμε ένα θησαυρό στην τσέπη και βγάζουμε τα χρήματα και τα διαθέτουμε ακόμα και εκεί που δεν είναι απαραίτητο. Γιατί λοιπόν δεν απευθύνουμε το ίδιο αίτημα και σε άλλους που έχουν το ίδιο καθήκον να υπερασπιστούν τόσο το στρατιωτικό σκέλος και την ειρήνη. Δεν πρόκειται εμείς να υπερψηφίσουμε την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να πω ότι έχουμε φαίνεται ένα πρόβλημα με τον όρο στρατιωτικός. Και θα δείτε και οι κλιματικές αλλαγές και η αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη θα μας οδηγήσει στην ανάγκη αντιμετώπιση κάποιων ε, κλιματικών αλλαγών ή συνεπειών των κλιματικών αλλαγών που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και οι συνέπειε δεν θα είναι τόσο στρατιωτικέ όσο ανθρωπιστικέ. Οπότε θα πρέπει να προσθέσουμε και το λόγο ανθρωπιστικό στο στρατιωτικό. Γιατί όταν έχουμε μία πλημμύρα ε, και θέλουμε να μετακινήσουμε πληθυσμό ε, μέσω των συστημάτων μεταφοράς, γιατί να προσθέσουμε και το ανθρωπιστικό στοιχείο εδώ. Επίσης, αυτά τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν θα πρέπει να εστιάζονται μόνο στο στρατιωτικό σκέλος. Γιατί με τις προσαρμογές που θα πρέπει να γίνουν θα εξυπηρετούν το σύνολο των μεταφορών. Προσοχή όμως, αυτά τα 6,5 δις είναι για τις μεταφορές, για την ε, ανακαίνιση των υποδομών, για την αύξηση της αστικής κινητικότητας. Έχουμε και εκεί σημαντικούς στόχους και θα πρέπει αυτούς τους στόχους να τους ε, χρηματοδοτήσουμε και με αυτή τη δημοσιονομική γραμμή, τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Κόλσον από την Γενική Διεύθυνση μου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ποιος είναι ο στόχος της πρότασης αυτής. Είναι η, να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει τις συνέργειες ή να αναδείξει κάποιες συνέργειες μεταξύ της πολιτικής μεταφορών και της αμυντικής πολιτικής. Και εγώ προσωπικά συμφωνώ μαζί σας. Προτιμώ τον όρο αμυντική πολιτική παρά στρατιωτικό, τον επίθετο στρατιωτικός. Γιατί όταν μιλούμε για αμυντική πολιτική έχουμε μια πιο ευρεία θεώρηση. Και έχετε απόλυτο δίκιο γιατί αυτές οι υποδομές θα εξυπηρετήσουν ε, εκφύσεως ε, και άλλους σκοπούς και όχι μόνο αμυγός στρατιωτικούς. Σίγουρα θα εξυπηρετήσουν, θα χρησιμοποιηθούν για σημαντικές μετακινήσεις, για ανθρωπιστικούς λόγους. Και ο στρατός στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζει και την πολιτική προστασία, οπότε θα χρειαστεί αυτές οι υποδομές και θα πρέπει να μπορεί να τις χρησιμοποιεί. Επίσης θα πρέπει να είμαστε σαφέστατοι εδώ. Ο μηχανισμός συνδέοντας την Ευρώπη σε καμία περίπτωση δεν θα χρηματοδοτήσει οτιδήποτε που δεν θα ε, εξυπηρετεί την πολιτική μεταφορών. Και στη δυτή χρήση έχουμε σαφή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να πραγματοποιήσει κάτι που ούτε θα χρειαστεί σε αμυντικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα θα είναι ωφέλιμο και για την πολιτική μεταφορών. Και αυτή η χρησιμότητα, αυτή η ωφέλεια θα ε, προσδιοριστεί με όλη την δέουσα διαφάνεια. Και θα επικοινωνήσουμε με τους ε, ενδιαφερόμενους των μεταφορών και θα τους ρωτήσουμε τι είδους επενδύσεις σε σχέση με τα κριτήρια που θα έχουμε προσδιορίσει σε στρατιωτικό επίπεδο θεωρούν ότι θα τους χρησιμεύσουν. Οπότε η τα κράτη-μέλη, οι ενδιαφερόμενοι για τις μεταφορές θα προσδιορίζουν τι είναι χρήσιμο για την πολιτική μεταφορά Και εδώ θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό θα μας επιτρέψει να κάνουμε κάτι περισσότερο για, το, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Γιατί από τη στιγμή που θα κρίνουμε ότι είναι κάτι χρήσιμο για την πολιτική μεταφορών, θα πρέπει κατά ανάγκη να συμπεριληφθεί στο, στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, στα TEN-T. Και στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, τα TEN-T, ε, θα χρηματοδοτήσουμε και το γενικό δίκτυο, που μέχρι στιγμής δεν έχουμε χρηματοδοτήσει αρκετά. Ή το κεντρικό δίκτυο, αλλά εκτός ε, διαδρόμων που μέχρι τώρα έχουν χρηματοδοτηθεί. Οπότε θα είναι αμοιβαίως ε, επωφέλης αυτή η προσέγγιση. Θα μπορούμε πιο γρήγορα να χρηματοδοτούμε χρήσιμα στοιχεία για τις μεταφορές στο σύνολο ε, του δικτύου των TNT, των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Επίσης, κάτι που δεν έχουμε χρηματοδοτήσει επαρκώς στο δικό δίκτυο στα πλαίσια του TNT. Εκεί θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε το συνδέοντα στην Ευρώπη ε, γιατί θα υπάρχει και στρατιωτικό ενδιαφέρον και ενδιαφέρον για τις μεταφορές. Οπότε, με την πρόταση αυτή θα είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι ε, στην πολιτική μεταφορών και θα έχουμε πολύ περισσότερα αποτελέσματα από ό,τι μέχρι στιγμής. Και τώρα, έρχομαι στο συγκεκριμένο σχέδιο, ε, στα συγκεκριμένα σχέδια. Η επιλογή των σχεδίων θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η επιλογή στα σχέδια του συνδέοντα στην Ευρώπη. Θα γίνεται διαγωνισμοί που ε, πρόκληση για την υποβολή προσφορών και θα, θα επιλέγουμε τα πιο ενδιαφέροντα, τα καλύτερα σχέδια. Και σίγουρα ο διασυνοριακό χαρακτήρα είναι σημαντικό κριτήριο. Γιατί το συνδέοντα στην Ευρώπη χρηματοδοτεί κυρίω διασυνοριακά σχέδια, άσχετα αν είναι χρήσιμα και για την αμυντική πολιτική. Και σίγουρα τα διασυνοριακά σχέδια θα έχουν προτεραιότητα στο συνδέοντα στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, σε καμία περίπτωση δεν θα αφαιρέσουμε προπολογισμό από το συνδέοντα στην Ευρώπη. Θα Μιλούμε εδώ για συμπληρωματικά κονδύλια και θα ως πρόσθετο προϋπολογισμός θα προτάθει κάτι τέτοιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν δούμε τις δημοσιονομικές προοπτικέ, βλέπουμε ότι το κονδύλιο αυτό είναι ξεχωριστό. Ε, είναι το κονδύλιο της αμυντική πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας. Και η διαχείριση αυτού του κονδυλίου θα γίνεται από το συνδέοντα στην Ευρώπη, από τη διευκόλυνση ΣΕΦ. Τώρα, για τα άλλα θέματα. Τίποτα δεν θα γίνεται αυθαίρετα. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διαδικασίες του μηχανισμού συνδέοντας την Ευρώπη. Αυτές οι διαδικασίες που τις γνωρίζετε θαυμάσια και που γενικώ δεν έχουν επισήρει επικρίσεις, αυτές οι διαδικασίες του συνδέοντας την Ευρώπη θα χρησιμοποιηθούν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κόλσον για τη διαφώτιση. Και τώρα ο εισηγητή μα πάλι, ο κύριο Τελίτσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και του συναδέλφους και όδης και όλους τους υπόλοιπους για τα σχόλιά σας. Συνολικά θα έλεγα ότι ήταν επί της ουσίας ε, οι παρατηρήσεις, πολύ εύστοχες. Και θα ξεκινήσω με το δικό σας σχόλιο, Πρόεδρε. Μιλήσατε για την ανθρωπιστική διάσταση. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή είναι καλή. Και είναι και κάτι που μπορούμε να το καλύψουμε. Νομίζω ότι και εσείς αυτό που, είπα, που είχα και εγώ κατά νου είπατε για στρατιωτικούς, πολιτικούς σκοπούς και επίγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες. Κάποιοι συνάδελφοι είπαν ότι θα καταψηφίσουν την πρόταση. Όμω, καλό θα ήταν να σκεφτείτε ότι σε κάθε κάτω μέρο μπορούμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου όταν υπάρχει φυσική καταστροφή ή κάτι κατασκευαστικό, ένα ατύχημα, θα πρέπει να κινητοποιηθεί ο στρατιωτικό εξοπλισμό και να μην επιτρέπεται ε, και ο κόσμο να βρεθεί σε κατάσταση απελπισία από την ε, καταστροφή και να μην μπορούμε να του βοηθήσουμε. Θα πεθαίνουν. Ε, λυπούμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ω προ την ανησυχία για τη δυτή χρήση θα μπορούσα να αναφέρω πολλά στοιχεία, πολλέ εκφράσει ε, του σχεδίου γνωμοδότηση, αλλά θα πω μόνο ένα παράδειγμα. Στην παράγραφο 5 θα πρέπει να είναι επιλέξιμο μόνο εάν προσθέτει κάτι σε υπάρχουσα υποδομή ή στο δίκτυο TNT, ώστε να μπορεί να υπάρξει διτή χρήση της υποδομής αυτής. Θα μπορούσα να δώσω πολλαπλά παραδείγματα, αλλά για μένα είναι ξεκάθαρο ότι η διτή χρήση είναι κάτι το πρόσθετο. Έρχεται ως κάτι το περαιτέρω. Και πρέπει να δούμε αν τα σχέδια, η σύλληψη των έργων, ε, η εκτέλεσή τους ε, μπορούν να ε, εξυπηρετήσουν σε αυτό το σκοπό. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πρόβλεψη έργου για αισθητοτικούς σκοπούς, ε, κυρίως ή αποκλειστικός. Ως προς τα χρηματοδοτικά μέσα που θα διαθέτουμε. Δεν ξέρω αν εδώ έχουμε την περίπτωση του αυγού με την κότα ή του μισοάδιου μισογεμάτου ποτηριού αλλά από τη σκοπιά του προπολογισμού ξέρω, δεν ξέρω μάλλον πώς κάποιοι φτάσαμε σε αυτό το συμπέρασμα. Η Επιτροπή προσθέτει ποσό. Δεν λέει κανείς ότι έχουμε 6,5 δις ε, ε, από μόνα τους χωρίς το χαρτοφυλάκιο. Λιγότερα θα είχαμε. Άρα δημιουργείται εδώ μια μορφή συνεργασίας, μια συνέργεια. Και το ποσό αυξάνεται και ο κύριος Φαντάλεν είπε κάτι που τον προβλημάτισε για το υποστηρίζουμε ε, στεναρός. Ε, λέμε, υποστηρίζουμε στεναρός την στρατηγική κινητικότητα στα πλαίσια της χρηστής διαχείρισης του προγράμματος ΣΕΦ. Αυτό λέμε. Σωστή διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Τώρα τι σας δυσκολεύει αυτό το strongly, το στεναρός. Ε, ε Καταρχήν λέτε ότι δεν συμφωνείτε με τη συμπερίληψη του στρατιωτικού χαρτοφυλακίου στο ΣΕΦ. Θέλετε να πάει αλλού. Δηλαδή να μην υπάρχει σχέση συνεργασίας και να χάσουμε και τη διετή χρήση που εδώ μπορούσαμε να επιδιώξουμε. Αυτό μας λέτε. Για τις τεχνικές ε, παραμέτρους. Βεβαίως δεν είναι μόνο τεχνικό το θέμα και σε κάποια θέματα θα μπορούσα να συμφωνήσω και με τον κύριο Φαντάλεν. Ναι, ε, εντάξει, πάντοτε όμως στην νομοθεσία έχουμε αυτή την προσέγγιση του σαλαμιού, ε, την προσέγγιση την κατατεμαχισμένη αναγκαστικά, γιατί μπορεί στο μέλλον να προκύψουν νέες εξελίξεις. Στην Ευρωπαϊκή Άμυνα μπορεί να προκύψουν νέες ανάγκες, αλλά αν δούμε το κείμενο προς στιγμήν, δεν καταλήγει στο να προτείνει μια συνολική έννοια τη Ευρωπαϊκή Άμυνα, παρόλο που εμένα θα μου άρεσε. Και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι ε, δεν ε, λέει κανείς ότι δεν θέλουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλουμε να κάνουμε οικονομίες. Και να το πω και να το ξαναπώ δεν θα απαγορεύσουμε στους εαυτούς μας να κοιτάξουμε τι γίνεται σε άλλες πολιτικές. Θέλουμε σχέση συνεργασίας, θέλουμε μείωση του κόστους και θέλουμε προστιθέμενη αξία. Νομίζω αυτά θα είχα να πω. Α, για, το, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα TNT. Χρησιμοποιήθηκε και άλλος όρος δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι πρόσθετο, αλλά με κάποιους διαδρόμους των δικτύων αυτών μπορεί να έχουμε μια νέα γραμμή και με μια αναβάθμιση να μπορεί κανείς, ας πούμε, σε μια συνδρομική γραμμή τρένου που έχει αντικατασταθεί από καινούρια, να πάρει την παλιά και να τη δώσει για στρατιωτικούς σκοπούς. Δεν θα επηρεάσει αυτό την υπόλοιπη κίνηση, την πολιτική, ας πούμε, συνδρομική γραμμή. Αλλά αυτό θα είναι μια εξαίρεση και είναι κάτι επιπλέον σε σχέση με αυτό που γίνεται τώρα. Αντί να σπαταλάμε χρήματα φτιάχνοντα μια καινούργια γραμμή από την αρχή, μπορεί να αξιοποιήσουμε την παλιά υποδομή. 6,5 δι είναι πολλά χρήματα, αλλά αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, θα βελτιώσουμε πολύ τι δυνατότητέ μα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Τελίτσκα. Και ευχαριστώ και του συναδέλφου για τη συζήτηση. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών λήγει την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου στι 5 το απόγευμα. Αυτή είναι η προθεσμία και να συνεχίσουμε με την κατεξουσιοδότηση πράξη για τα ευφύ συνεργατικά συστήματα μεταφορών. Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα εγκρίνεται σύντομα κατεξουσιοδότηση πράξη για τα ευφυή συστήματα, τα συνεργατικά συστήματα μεταφορών, τα γνωστά και ως SITS. Η CETS. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Σουγέλη και την ε, κατεξοδότηση πράξη θα την λάβει επισήμως στο Κοινοβούλιο ε, Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Να δώσω το λόγο στον κύριο Βαντίλεν. Ε, πού είστε, ε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Και υπενθυμίζω καταρχάς τι συζητούμε εδώ. Καταρχάς έχουμε να κάνουμε με στόχους μεταφορών, περιορισμό των ε, ε, συμφορήσεων, ε, άνοιγμα των μεταφορών προς όλους, ενίσχυση βέβαια και της ηγετικής θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε επεξεργαστεί διάφορα στοιχεία, διάφορες συνιστώσεις, πλατφόρμες, πολιτικές, υπερσυνοριακά έργα και έργα μεγάλης κλίμακας. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν είναι το πρώτο βήμα μόνο, πρέπει να το εξηγήσω, δηλαδή σύνδεση οχημάτων που μπορούν έτσι να επικοινωνούν μεταξύ τους, να συνεργάζονται και να καθιστούν πιο ασφαλείς τις μεταφορές. Ένα όμως μόνο πρώτο βήμα ως προς την υψηλή αυτοματοποίηση, όπου αναμένεται εν τέλει να μπορούν όλα τα οχήματα να συντονίζουν τις κινήσεις τους και να εξασφαλίσουμε μηδενικό ατύχημα, μηδενικό θάνατο στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Κάτι εξουσιοδότηση πράξη λοιπόν, ως τελευταίο βήμα τεσσάρων διαφορετικών στοιχείων, γιατί ξεκίνησαμε με ένα κοινό όραμα, με την ε, συζήτηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, ενδιαφερομένων παραγόντων, βιομηχανίας, ε, κρατών κτλ. Μετά έχουμε τα μεγάλα έργα μεγάλης κλίμακας με 16 κράτη-μέλη σε πλήρη ανάπτυξη και άλλα τέσσερα σε παρακολούθηση των συνομιλιών. Και τώρα το τελευταίο αυτό κομματάκι του μοσαϊκού είναι το, η κατεξουδότηση στην πράξη. 16 κράτη-μέλη είπα ήδη έχουν αναπτύξει προγράμματα, βεβαίως σε συνεργασία και με, την, ε, με τον κλάδο, με αρκετούς μεγάλους παράγοντες του κλάδου που συμμετέχουν και είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στην ανάπτυξη, γιατί το CATS σημαίνει αφενός μεν υποδομές, επικοινωνία δηλαδή με τα οχήματα, αλλά η μεγαλύτερη επένδυση και το κόστος θα έχει να κάνει με τον εξοπλισμό όλων των οχημάτων όταν έρθει η ώρα. Και εδώ πάλι έχουμε πολλή υποστήριξη και πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε. Πρόκειται και μια ιστορία που έχει πίσω τις 10 χρόνια συζήτησης και προσπάθειας. Ήδη προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε το CATS νωρίτερα. Δεν τα καταφέραμε. Ελπίζουμε ότι τώρα είναι δυνατόν ε, για να τα καταφέρουμε όμως χρειαζόμαστε τη βεβαιότητα που μπορεί να προσφέρει ε, το νομοθέτημα. Μπορώ να σας δώσω και λεπτομέρειες του νομοθετήματος του ίδιου, αν σας ενδιαφέρει, αλλά για να κερδίσουμε χρόνο θα προτιμούσα να ακούσω τις ερωτήσεις σας για να απαντήσω συγκεκριμένα. <coughs> Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κάμπ, έχετε ζητήσει πρώτο το λόγο, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι καταλαβαίνει τα δικά ο κύριος τη επιτροπή, οπότε θα είναι πιο εύκολα. Στο ΕΛΚ λοιπόν. Έχουμε κάποιες επιφυλάξεις σχέση με τις κατεξουσιοδότητες πράξεις. Και πιστεύουμε ότι πρέπει με προσοχή να εξετάσουμε το θέμα. Και τα αισθήματα είναι τα εξής. Πρώτον, πώς θα υλοποιηθεί η κατεξουδότηση πράξη, εάν δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιο είναι ο γενικό κανονισμός για την προστασία των δεδομένων, τη λειτουργία του και τον αντίκτυπο που θα φέρει. Ποια θα είναι η λειτουργία του και ο αντίκτυπο που θα φέρει, αφού ακόμα ίσα ίσα έχει αρχίσει να τεθεί σε εφαρμογή. Επομένω, τι συνέπειε θα έχει αυτό για το CITS. Δεν πρέπει να περιμένουμε πρώτα αυτό. Επίσης για την Επιτροπή οι τεχνικές εξελίξεις φαίνεται να προχωρούν ταχύτερα από ότι η εξέλιξη της κατεξουσιοδότησης πράξης. Η τεχνολογία 5G θα ενσωματωθεί λοιπόν στην κατεξουσιοδότηση πράξη. Αφού ήδη χρησιμοποιείται με την εξέλιξη τεχνολογία στα οχήματα, προβλέπετε κάτι τέτοιο. Το έχει υπόψη η Επιτροπή. Εδώ έχουμε να κάνουμε όχι μόνο με την αυτοκινητοβιομηχανία εννοείται, αλλά και με άλλους τομείς. Επίσης, γενικός κανονισμός για την ασφάλεια, προστασία δεδομένων, αλλά και γενικά η ασφάλεια. Τι δράση, τι αλληλεπίδραση βλέπουμε μεταξύ αυτού του νομοθετήματος και της κατεξουδότησης πράξης. Μετά, βιομηχανία και κράτη-μέλη. Λέτε ότι συμμετέχουν στην εξέλιξη της κατεξουδότησης συμπράξης. Πώς? Πολύ να μας λέει η Επιτροπή ότι του ακούει, έχει την ευήκονους λοιπά Ναι, αλλά πέραν του να ακούμε πρέπει και να δρούμε, δηλαδή να προσαρμόζουμε το νομοθέτημα σε αυτό που μας έχουν πει. Μετά, ε, μελέτη αξιολόγησης έχει προβλεφθεί ή αντικτύπου θα γίνει διαβούλευση δημόσια. Πώς θα διαμορφωθεί αυτή. Με τι διατυπώσεις. Αυτοκίνητο βιομηχανία. Επηρεάζει ή όχι. Κύριε Βαντενκάμπ. Ευχαριστώ κύριε Βαντενκάμπ. Έχετε το λογο Ε, βρείτε τα μεταξύ σας λοιπόν. Οποιο είναι να ξεκινήσει. Κύριε Ερτούγα, εσεί. Ευχαριστώ. Ο Ιστβάν είναι ο εισηγητή και θα πει πολύ περισσότερο από ό,τι εγώ, αλλά ε, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι. Καταρχά, να ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βεβαίω. Ε, με όλες τις επικρίσεις βλέπουμε ότι έχει επιληφθεί και έχει διαμορφώσει τις προτάσεις Πριν από ένα χρόνο είχαμε απορρίψει και επικρίνει πάρα πολλά πράγματα και βλέπουμε ότι έχει σχετικά προσαρμοστεί. Υπάρχουν και ειδικοί, υπάρχουν οι ομάδες των εμπειρογνωμόνων ε, και σε επίπεδο βέβαια επιτροπής έχει γίνει επεξεργασία των θεμάτων. Έστω πολύ αργά δυστυχώ, αλλά έστω. Αυτό λοιπόν που με ενδιαφέρει είναι πρώτον γιατί το κάνουμε αυτό. Θέλουμε στο μέλλον να έχουμε αυτοματοποιημένη και ε, ενοποιημένη, ε, συνδεδεμένη κινητικότητα, πράγμα το οποίο θα μας ε, επιτρέψει να αποφύγουμε και ατυχήματα και κυκλοφοριακές συμφορήσεις και πολλά άλλα. Και επιπλέον πώς μπορούμε σε μια Ευρώπη των 28 κρατών μελών να υλοποιήσουμε αυτή την συνδεδεμένη κινητικότητα. Εδώ λοιπόν η ανησυχία η δική μου είναι ότι πολλές φορές στις Βρυξέλλες μαζεύουμε, συγκεντρώνουμε όλη αυτή την τεχνογνωσία, τις προτάσεις, τις ιδέες και μετά όταν έρθει η ώρα της υλοποίησης εξαρτώμεθα από το κατά πόσον θα συμπράξουν τα κράτη-μέλη. Ε, και στρέφοντας το βλέμμα προς τα κράτη-μέλη, τα επιμέρους, βλέπω ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικά επίπεδα σε υποδομές, και θα το πω ε, κάπως διπλωματικά και ορίμανση σε επίπεδα διαφορετικά, ορίμανση τόσο σε νοοτροπίες ε, πολιτισμικά δηλαδή, αλλά και σε υποδομές. Πώς λοιπόν μπορούμε να εξασφαλίσουμε, η Επιτροπή δηλαδή, πώς θα εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη θα κάνουν αυτό που οφείλουν και μάλιστα σε ένα ε, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ορατό χρονικό διάστημα πριν καταστεί και επικίνδυνη η κατάσταση, γιατί ξεκινάει η αυτόνομη οδήγηση, είτε το θέλουμε είτε όχι. Και επίσης για να ε, πιαστώ και από τα λόγια του κυρίου Φαντενκάμπ. Πολλοί λένε ότι μπορεί το Wi-Fi να είναι ένα σύστημα ε, στεναρό, γερό, που μπορεί να χρησιμοποιείται μεν, αλλά δεν είναι επαρκές για τις τεχνολογικές εξελίξεις και υποστηρίζουν ότι πρέπει να προχωρήσουμε αμέσως στο 5G, στο 5G. Γιατί λοιπόν αυτό το έχει αποκλείσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί να μην προσπαθήσουμε να το ενσωματώσουμε στις οδικές μας υποδομές. Γιατί δηλαδή να επενδύσουμε σε μια τεχνολογία που ήδη την έχει ξεπεράσει κάτι άλλο πολύ καλύτερο. Ή, εν πάση περιπτώσει, για να μην χρησιμοποιώ τη λέξη καλύτερο εύκολα, ας μου εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι είδους επιφυλάξεις μπορεί να έχει έναντι της τεχνολογίας 5G. Ευχαριστώ. Πρέπει να επιταχύνουμε λίγο τώρα τους ρυθμούς μας, γιατί μένουμε όλο και πιο πίσω. Κύριο Στελίτσκα. Κύριε Πρόεδρε, καλώς. Τότε να είμαι πολύ λακωνικός εκπροσωπώ την κυρία Μάισνερ που δυστυχώς είχε κάποιο πρόβλημα υγείας και τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά παρακολουθεί το ζήτημα πολύ στενά και δεν έχει ιδιαίτερες ανησυχίες ή προβλήματα. Θεωρούμε ότι έχει σημειωθεί εντυπωσιακή πρόοδος που ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες της Επιτροπής Μεταφορών. Το μόνο σημείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι κάτι που ήδη αναφέρθηκε Οπότε δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Είναι το θέμα του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, GDPR. Νομίζω ότι ε, οι φιλελεύθεροι μπορούν να μείνουν ικανοποιημένοι από τα πραγμένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Ουλέλη, πολύ σύντομα όμως παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε. ότι az elmult ε, θα ήθελα λοιπόν και εγώ να επισημανώ ότι κάπως με εξαφνιάζει το πόσες οργανώσεις επαγγελματιών με έχουν προσεγγίσει, έχοντας αναλάβει την έκθεση CATS, ε, νομίζω ότι μπορώ να γνωρίζω τα πράγματα καλά. Υπάρχει ένα συντονισμός, αλλά φαίνεται να έχουν ξεσηκωθεί οι επαγγελματίες όπως είχε γίνει με την έκθεση ITS, αν θυμάστε. όπου με την εμφάνισή της ε, προκλήθηκε μεγάλος δώρος και αναστάτωση και μετά κάπως ηρεμήσαν τα πνεύματα. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε έγκαιρος, ώστε δυνατόν πιο νωρίς να έρθει σε επαφή και να επικοινωνήσει με τις οργανώσεις των επαγγελματιών, ώστε να μην υπάρξουν ε, αναταραχές χωρίς λόγο. Έχουμε πολλά θέματα να επεξεργαστούμε πάνω στο νέο σύστημα, αλλά πρέπει να ακούσουμε πάνω απ' όλα τις οργανώσεις, εκείνους που ξέρουν το πράγμα από τη δουλειά τους. Το Wi-Fi επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ε, ή μάλλον συγγνώμη, ο κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πολύ μεγάλη σημασία και το πώ θα συνδυαστεί με το CITS. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε κάποια στιγμή, στοιχεία που να μα δείχνουν ότι, συγκερα... ότι μπορούμε να συγκεράσουμε τα μελήματα των μεν και των δε. Σα ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση μόνο για τις έξυπνες συνεργατικές μεταφορές. Μας είπατε στην ομιλία σας ότι θα ήθελατε να, γίνει, να έχει γίνει πιο νωρί η ανάπτυξή του. Πάει μια δεκαετία που ασχολείστε με το θέμα αυτό. Πώ εξηγείται αυτή την καθυστέρηση, γιατί δεν μπορούμε επιτέλου να περάσουμε στη φάση τη ανάπτυξη, Ποια είναι τα προσκόμματα, τι μα έχει εμποδίσει μέχρι στιγμή να προχωρήσουμε. Γιατί αυτό είπατε, ότι θα, ήθετε, θα θέλατε να είχατε προβεί στην ανάπτυξη πολύ πιο νωρί. και ότι εδώ και 10 χρόνια ασχολείστε με το θέμα αυτών των έξυπνων συνεργατικών μεταφορών. Οπότε η ερώτηση μου είναι απλή. Ποια είναι τα προσκόμματα στα οποία προσκρούσατε, γιατί δεν έγινε μέχρι στιγμή η ανάπτυξη και έχετε καθυστερήσει τόσο πολύ. Ο λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Βαντερλίντα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ εύστοχε οι ερωτήσει σα. Ξεκινώ από την τελευταία, τη δική σα, Γιατί χρειάστηκε να περάσει μια δεκαετία. Όταν είπα 10 χρόνια, ενώ οπότε ξεκίνησε η έρευνα. Η έρευνα όντω ξεκίνησε πριν από 10 περίπου χρόνια. Και η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονό ότι πρόκειται για ένα θέμα που προϋποθέτει συνένεση των πάντων για το ίδιο θέμα. Ε, δεν μπορούμε να περάσουμε στη φάση της ανάπτυξης και της εφαρμογής αν δεν έχουμε πλήρη εκτεταμένη συνεννόηση και συμφωνία, ολόκληρο κλάδων. Και απαιτείται πλήρη συμφωνία, κάτι που δυσκολεύει τα πράγματα. Δεύτερον, παρόλο που κανένα δεν αφιβάλλει για τα κοινωνικά ωφέλη των έξυπνων συνεργατικών μεταφορών, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα κοινωνικά πλέον εκτήματα, όλοι θα βγουν κερδισμένοι, αλλά το θέμα είναι ποιο θα βγάλει χρήματα, ποιο θα βγει ο πιο κερδισμένο. Θα πρέπει λοιπόν να μεταφέρουμε και σε καλό επιχειρηματικό μοντέλο αυτά τα κοινωνικά ωφέλη. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τους καλούς λόγους και τα κίνητρα για να μπορέσουν να επενδύσουν. Και αυτό είναι δύσκολο να το βρούμε και χρειάζεται χρόνος, είναι χρονοβόρα διαδικασία. Για να γίνουν οι αλλαγές λοιπόν, χρειάστηκε εκτεταμένη συνεννόηση με όλους τους εφεροντούχους και με τον κλάδο. Γιατί όπως είπα, οι μεγαλύτερες επενδύσεις θα γίνουν από τον κλάδο, από τον εξοπλισμό των οχημάτων. Οπότε δεν είχαμε επαφέ με την βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία, δεν είναι πρόκειτο να περάσουμε στην φάση τη έμπρακτη εφαρμογή. Στο μεταξύ έχουμε προσυδεριστεί τη βιομηχανία και πολλοί ενδιαφερόμενοι ε, και κατασκευαστέ ε, ε, έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους επίσης και οι κατασκευαστές μοτοσυκλετών έχουν εκφράσει ενδιαφέρον. Έχουμε τη δέσμευση 16 κρατών μελών που έχουν στενή συνεργασία και κοινή ανάπτυξη με τον κλάδο, με τη βιομηχανία. Γι' αυτό έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή θα περάσουμε επιτέλους στην πράξη. Πολλοί εξέφρασαν ε, ανησυχίε για το Γενικό Κανονισμό προστασία Δεδομένων. Φυσικά ο GDPR είναι εφαρμοστή νομοθεσία και η καταξιοδότηση πράξη δεν, πρέπει να αλλάξει, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι τέτοιο, ούτε να ερμηνεύσει τον κανονισμό για την προστασία δεδομένων. Απλώ θα αλλάξουμε κάποια πρακτικά θέματα. Και στην πράξη ελάχιστα μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτοί που θα ε, προβούν στην ανάπτυξη ε, και ο τρόπο με τον οποίο θα κάνουν την ανάπτυξη προποθέτει. Ε, προηγούμενη απόδειξη ότι οι δράσεις τους ευθυγραμμίζονται με το GDPR. Αυτό είναι ε, φυσικά αρμοδιότητα των αρχών προστασίας δεδομένων. Πολλοί αναφέρθηκαν και στις νέες τεχνολογίες. Εκτιμούμε ιδιαίτερως αυτό το σχόλιο. Και θα πρέπει να είμαστε όσο πιο ανοιχτοί γίνεται στις νέες εξελίξεις. Και η καταξιδότηση πράξη το αναφέρει ρητά. Γιατί αυτή είναι η στρατηγική μας, ότι δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. 26.000 άνθρωποι αφήνουν τη ζωή τους στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Θα πρέπει λοιπόν το συντομότερο δυνατόν να ανταποκριθούμε και να μειώσουμε αυτά τα τροχέα με τις τεχνολογίες που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, αλλά να είμαστε ανοιχτοί και στις μελλοντικέ τεχνολογίες. Και η καταξιοδότηση πράξη προβλέπει ρητά ότι στο μεταξύ που θα είναι έτοιμες νέε τεχνολογίε για ανάπτυξη και με έναν αρμονισμένο τρόπο θα γίνει αναθεώρηση της κατεξοδότηση πράξης. Δεν θα περιμένουμε μία άλλη τριετία ή πενταετία για να συμπεριλάβουμε τις νέες τεχνολογίες. Και τέλο, μελέτη επιπτώσεων. Αυτή εκπονείται εκ παραλίλου και θα είναι έτοιμη μαζί με την κατεξοδότηση πράξη. Ελπίζω να απάντησε στι απορίε σα και μάλιστα εγκαίρως. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βαντερλίνε. Κύριε Βίμ Βαντερκάμ, παρακαλώ όμω πάρα πολύ σύντομα γιατί περι... μας περιμένει ο κύριο Ολολέη. Κύριε... Κυρία Πρόεδρε, ε, ήθελα απλώς ε, να μας κάνετε τη σύνδεση με το γενικό κανονισμό για την ασφάλεια. Ναι, όντως, ε, πολύ εύστοχη ερώτηση, το ξέχασα. Όπως δείχνει και η οθόνη, είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι η συνδεσιμότητα, τα συνεργατικά συστήματα και τα αυτοματοποιημένα συστήματα θα πρέπει να συγκλίνουν. Αυτά είναι τα τρία συστήματα που μέχρι στιγμής είχαν αναπτυχθεί ξεχωριστά και πιστεύουμε ότι θα πρέπει επιτέλους ε, να συμβαδίζουν, να συγκλίνουν. Ήδη έχουμε διερευνήσει πολλές συνέργειες και έχουμε ε, ανακοίνωση ώστε να μπει η έξυπνη συνεργατική μεταφορά στη, στο τρίτο πακέτο για την κινητικότητα ε, και την συνδεσιμότητα. Θέλουμε να ε, αξιοποιήσουμε τα ωφέλη όλων αυτών των συνεργειών. Τα συστήματα είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους και όλα τα συστήματα αυτά είναι χρήσιμα και απαραίτητα. Σε ευχαριστούμε κύριε Βαντελίντε ε, για την ανταλλαγή απόψεων και σίγουρα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό και στο μέλλον. Περνάμε τώρα... Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρησης διάταξης, την ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Διευθυντή της ΜΟΥΦ, τον κύριο Ολολέη. Η τελευταία μας ανταλλαγή απόψεων έγινε το Σεπτέμβριο του 2017, δηλαδή πριν από ένα χρόνο, οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε τον επωφελή διάλογο για τα δύο θεσμικά όργανα και άλλωστε δεν θα περιοριστούμε μόνο στο πακέτο για την κινητικότητα. Έχουμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων προ συζήτηση και ευχαριστούμε τον κύριο Ολολέη που ήρθε στην Επιτροπή για να μα παρουσιάσει τι προτεραιότητε Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλου του κλάδου των μεταφορών θα μας κάνει και έναν απολογισμό των αποτελεσμάτων και μία παρήθμιση των προκλήσεων που θα πρέπει από κοινού να αντιμετωπίσουμε μέχρι το πέρας της κοινοβουλευτικής μας θητείας και φυσικά και επέκεινα, αλλά και σίγουρα μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας, δηλαδή για το επόμενο οκτάμινο. Μετά την ομιλία του κ. Λολέη θα γίνει συζήτηση με τους συντονιστές και τους υπόλοιπους βουλευτές. Κύριε Λολέη, έχετε το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητή Καρίμα, κυρίες και κύριοι, βουλευτές και μη. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι και πάλι εδώ στην Επιτροπή ΤΡΑΝ για την σημερινή μας συζήτηση. Δεν σας έχει διαφύγει το γεγονός ότι ο χρόνος τρέχει. Είμαστε στι τελευταίε φάσει αυτή τη θητεία του Ευρωκοινοβουλίου και τη Επιτροπή Γιούνκερ. Θέλω λοιπόν να τονίσω πως έχω εκτιμήσει την αφοσίωση, βαθιά εκτίμησα την αφοσίωσή σα, στην ε, πρόοδο που θελήσατε να επιτελέσουν ε, οι μεταφορέ και οι πολιτικές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής. Και επίσης εκτίμησα ιδιαίτερα την ε, στενή μας συνεργασία είναι θέμα, είναι θέμα αποφασιστικότητας και εργατικότητας για να πετύχουμε κοινούς στόχους. Είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε, πετύχαμε αρκετά και θα πετύχουμε και άλλα στο μέλλον. Ευχαριστώ όλους για τη συμβολή σας σε μείζονο σημασία εκδηλώσεις που οργάνωσαν, στήριξαν και οι υπηρεσίε της Επιτροπής, όπως το άτυπο Συμβούλιο του Τάλιν τον περασμένο Σεπτέμβριο, τη συνδιάσκεψη για τη σύνδεση της Ευρώπης, εκεί όπου καλήσαμε για ενίσχυση του ΣΕΦ στο επόμενο πουδουπού και επίσης την ε, συμμετοχή σας στις ημέρες TNT στη Λιουμπλιάνα. Με την εξαιρετική σας στήριξη υπογραμμίσατε την πολιτική διάσταση της δουλειάς μας στις μεταφορές. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ ειλικρινά. Και αυτό ισχύει για πολλά μέλη της Επιτροπής σας, αλλά όλος ιδιαίτερος για την πρόεδρό της, την Καρή Μαντελή, της οποίας η συμμετοχή και οι σκόπιμες παρεμβάσεις, καθώς και η διάθεση να είναι επικοδομητική, ήταν κλειδί για την επιτυχία αυτών των εκδηλώσεων και για τη συνεργασία μας εν γέννη. Επειδή βρισκόμαστε στα τελικά στάδια τη συνεργασία μα κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία, νομίζω καλή ευκαιρία θα ήταν σήμερα να, πάρουμε, να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να σκεφτούμε και να παρατηρήσουμε τι πετύχαμε από κοινού. Όμω, εξίσου σημαντικό είναι να σφιγμομετρήσουμε λίγο την πρόοδο στα θέματα που βρίσκονται ακόμη στο τραπέζι των δημοτεύσεων, γιατί έχουμε λίγο αλλά πολύτιμο χρόνο για να πετύχουμε πρόοδο ακόμη και τώρα. Οι μεταφορές έχουν να αντιμετωπίσουν ε, ε, προβλήματα άνευ προηγουμένου, αλλά και μοναδικέ ευκαιρίε, απειλέ ασφάλεια, προβλήματα στην ψηφιοποίηση, απαλλαγή από τον άνθρακα και την αλλαγή στα επιχειρηματικά μοντέλα τη παγκοσμιοποίηση. Θα πρέπει λοιπόν με θετικό τρόπο να βρούμε λύσει για αυτά τα προβλήματα και με προτάσει πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο, για να πετύχουμε και άλλε επιτυχίε. Ποια είναι τα βασικά μα επιτεύγματα. Να αναφέρω μερικά. Γενικώ, τα θέματα μεταφορών μπήκαν λίγο στο επίκεντρο της προσοχής του κοινού ε, τα προβάλαμε μαζί με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων ε, ποιοτικών θέσεων εργασίας. Η επιτυχία της προσέγγισης αυτή αυτής φάνηκε και με, το, ε, με την διευκόλυνση για την διασύνδεση της Ευρώπης και με άλλα κονδύλια που ίσως να ληφθούν υπόψη για την πρόοδο των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με, το, με τις προτάσεις μας για τη δυτή κινητικότητα μπορούμε να πετύχουμε μια βιωσιμότερη διαχείριση των μεταφορών από ό,τι στο παρελθόν. Στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι μεταφορές είναι μια σημαντική και απαραίτητη συνιστόσα. Ω προ τα συγκεκριμένα θέματα, πριν από λίγο καιρό, και θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σα, μας στηρίξατε για, την, για να εγκριθεί το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο στα τέλη του 2016, καθώ και κατά εξουσιοδότηση πράξη για, την, για ε, τον προγραμματισμό των έργων υποδομών μέχρι το τέλο του 2017. Επιπλέον, η Επιτροπή Τραν ασχολήθηκε και εργάστηκε ε, εντατικά για να πετύχουμε θετική συμφωνία στο νέο βασικό κανονισμό για την ΕΑΖΑ. Ο κανονισμό αυτό θα τεθεί σε ισχύ σε λιγότερα από μια εβδομάδα. Γι' αυτό θέλω να υπογραμμίσω το ζωτικό ρόλο του Κοινοβουλίου στην ε, αλλαγή τη πρόταση, τη αρχική πρόταση με τι πολύτιμε τροπολογίε του. Ιδίω τον κύριο Μαρινέσκου, τον εισηγητή, του οποίου η αμέριστη στήριξη ήταν ε, μεγάλη σημασία για να πετύχουμε ένα ισορρόπο αποτέλεσμα και στο Συμβούλιο. Ο κανονισμό θα διασφαλίσει ασφαλή ε, περιβαλλοντικώς φιλικά ε, συστήματα αεροπλοείας για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ε, καλύψει κενά στο ρυθμιστικό σύστημα με αποτελεσματικό σύστημα ε, ασφάλειας και διαχείριση της ασφάλειας και τη σχετική συνεργασία και με νέα τεχνολογικά μέσα. Το ίδιο και με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη ασχέτως του βάρου Βάρους τους. Έτσι θα γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στο παγκόσμιο προσκήνιο. Στι χρυσέ μεταφορέ ξέρω ότι η οδική ασφάλεια είναι από τι πρώτε σα προτεραιότητε, όπω και για μα. Γι' αυτό λοιπόν ε, θέλω να σα ευχαριστήσω για την ε, στεναρή σα στήριξη την διαρκή σα στήριξη στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Η ταχεία έγκριση και η βελτίωση τη πρότασή μα για τα επαγγελματικά προσόντα των επαγγελματιών οδηγών ήταν μια κοινή επιτυχία. Όμω μπορούν να γίνουν περισσότερα και εδώ. Και υπάρχει, ήταν σημαντική η συμφωνία για την ε, αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τη εσωτερική των ε, πιλότων στην εσωτερική πλοία μέχρι το τέλο του 2017. Είναι σημαντικό και αυτά τα επαγγέλματα να γίνουν πιο ελκυστικά. Γι' αυτό λοιπόν η αυξημένη προσοχή της τραν στα θέματα αυτά ήταν για μας ε, πολύ σημαντική για τις προκλήσεις που απομένουν. Ε, μερικά παραδείγματα για το τι σημαντικό έχουμε πετύχει από κοινού έδωσα μόλις τώρα. Να περάσω τώρα στο τι έχουμε μπροστά μας τους ερχόμενους μήνες. Και είναι πολλά. Ε, ο μακροπρόθεσμος, ο πολιετής προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπός Μπούλτ και οι επιτηρησίε μας υπέβαλαν πρόταση για το ΣΕΦ για το 2021-2027 και τα έχετε δει αυτά που προτείναμε. Χαιρόμαστε που η Επιτροπή σα έχει προετοιμάσει ήδη την πρώτη εξέταση του σχεδίου αυτού. Για το ΣΕΦ 2 θα είναι ζωτική σημασία να έχουμε ταχεία πρόοδο για να είμαστε βέβαιοι ότι το νέο πλαίσιο για τη χρηματοδότηση θα εγκριθεί πριν το τέλο αυτή τη κοινοβουλευτική θητεία. Ε, Προλαμβάνοντα την λήξη τη προθεσμία για την αποβολή των πολεμιών, να επαναλάβω τα εξή. Για την περιοδο 2021 2021-2027 εκτιμούμε ότι το βασικό δίκτυο του TNT θα πρέπει να υπερκοδοτηθεί με 350 δι επενδύσει και επιπλέον 700 δι για το συνολικό δίκτυο και τι ανάγκε μεταφορών. Δεδομένων αυτών των επενδυτικών αναγκών, προτείναμε ενισχυμένο ΣΕΦ με ένα συνολικό προπολογισμό 42,3 δι, εκ των οποίων 30,6 δι ε, ε, θα κατευθυνθούν τι μεταφορέ. Η πρότασή μας είναι και για το Γενικό Χαρτοφυλάκιο και για το Χαρτοφυλάκιο Συνοχή ε, στο πλαίσιο του Πουδουπού. 12,8 δι και 11,3 δι αντιστοίχω. Επιπλέον, ε, στην ε, στρατιωτική κινητικότητα βρισκόμαστε πλέον σε νέο επίπεδο. Με την με το δίκτυο, με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, το TNT, να είναι μοχλό για να προχωρήσουν σε θετικέ και πολιτικέ ανάγκε των μεταφορών ε, και να καλύφθουν ταυτόχρονα. Επίση, πρόσφατα δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα εργασιών των Ευρωπαίων Συντονιστών από το TNT, με συγκεκριμένου βασικού ε, διαδρόμους διασύνδεση και τα λεγόμενα ERTMS, με τους ε, αυτοκινητοδρόμου τη θάλασσα, τις λεωφόρου τη θάλασσα. Θα πρέπει αυτού του στόχου να του επιδιώξουμε στο 2030, αλλά και μετά το 2013 ο κανονισμό ε, του TNT, όπω τον έχουν μελετήσει στα τέσσερα τελευταία χρόνια οι Ευρωπαίοι συντονιστέ θα πρέπει να προχωρήσει. Ε, οργανώσαμε σχετικά ακροάσει και στην Επιτροπή και στη δική σα Επιτροπή. Και είμαστε βέβαιοι ότι οι μελλοντικοί ε, Ευρωπαίοι συντονιστέ, η κυρία Ραντίτσοβα Γένσεν και ο κύριο Ρούτε, θα αναλάβουν με επιτυχία τη θητεία του και θα ενισχύσουν την ομάδα των συντονιστών. Σε συνδυασμό με το ΣΕΦ, προτείναμε και ένα σχέδιο κανονισμού για να ευθυγραμμίσουμε τι διοικητικέ διαδικασίε και να διευκολυνθεί η υλοποίηση των έργων TNT. Στόχο είναι να βελτιώσουμε και να προσφέρουμε μεγαλύτερη σαφήνεια στην εκτέλεση των προγραμμάτων καθώς και να μειώσουμε το κόστος. Από το 2014 ε, ε, υποστηρίξαμε πάνω από 640 έργα με κόστος ε, πάνω από 23 δι. Συνολικέ επενδύσει 45 δι ευρώ. Αυτό αφορούσε τουλάχιστον 2.000 δικαιούχους ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προγράμματα αυτά σκοπό είχαν τη βιώσιμη ανάπταξη των ε, μεταφορών, των σιδηροδρόμων και τη εσωτερική ναυλοπλοεία, καθώ και άλλε προτεραιότητε όπω την κοινοτομία και τα τεχνολογικά συστήματα, για την ε, ενίσχυση τη ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα. Ε, γι' αυτό τα 23 δι που προέβλεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύτηκαν αμέσω στην πρώτη τριετία λειτουργία του ΣΕΦ. Αυτό σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και συνεχίζουμε να προωθούμε το ΣΕΦ με τρόπο δραστήριο. Πολύ σύντομα θα διατεθεί όλο το ποσό. Οι σχετικοί διαγωνισμοί θα ανακοινωθούν σύντομα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ίδιο και η διαδικασία ε, για το 2018, το διαγωνισμό των φετινό, με υποβολή προτάσεων στα τέλη Οκτωβρίου και την επιλογή στι αρχέ του επόμενου χρόνου. Ε, ψηφιοποίηση, οδική ασφάλεια και ε, τη χρήση θα είναι μερικά από τα θέματα που μας, ε, θα μα απασχολήσουν του χρόνου. Και το 2019 θα έχουμε ένα διασυνοριακό έργο για το συνολικό δίκτυο και την ηχορύπανση που πρότεινε η Επιτροπή σα. Ω συνήθω, είμαστε στη διάθεσή σα για να ενημερώσουμε για τι πρωτοβουλίε και τα επόμενα βήματα. Να περάσω τώρα στα πακέτα διδέσμιου μέτρων για την κινητικότητα. Οι προτάσεις αυτές παρουσιάστηκαν πρόσφατα. Τα σημαντικά αυτά πακέτα επιβεβαιώνουν την προτεραιότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να ολοκληρώσει και να εξυγχρονίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις μεταφορές και υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Εάν δεν πετύχουμε πρόοδο στα θέματα αυτά, θα έχουμε χάσει μια ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώ. Για την πρώτη δεσμή μέτρων για την κινητικότητα. Ξέρετε ότι οι προτάσει μα συνεχίζουν να διχάζουν. Όμω ευτυχώ έχουμε πετύχει πρόοδο σε πολλά θέματα. Γι' αυτό καλωσορίζω την έναρξη των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο. Με τον πρώτο τριμερή διάλογο να γίνεται στις 11 Ιουλίου φέτος. Είναι ένας τεχνικός φάκελος, ένα τεχνικό θέμα αυτό που ελπίζουμε να ολοκληρωθεί εγκαίρως. Επίσης χαίρομαι που το Κοινοβούλιο ψήφισε την εκθεσή της για τα ΕΦΗ δίκτυα, αν και το Συμβούλιο δεν έχει πετύχει ακόμα μια προσέγγιση. Καταλαβαίνω ότι οι δημοτεύσεις για το φάκελο αυτό είναι πολλαπλές και έχουν να κάνουν με άλλες δημοτεύσεις για την εσωτερική αγορά. Δεν βλέπω όμως να υπάρχουν φοβερές διαφωνίες για τη συνολική μας προσέγγιση ούτε στο Συμβούλιο ούτε στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ όλους τους εισηγητές ε, της Επιτροπής Τραν, ε, Σαλίνη Μοντέρο, ε, για τα πακέτα κινητικότητας και την ε, συνεισφορά σας. Γιατί και στον κοινωνικό πυλώνα και τον πυλώνα της εσωτερικής αγοράς μας ενισχύσατε και στο θέματα του καμποτάζ και σε πολλά άλλα. Ευχαριστώ και τους κοιόδης εισηγητές για την εντατική τους δουλειά. Ωστόσο, είναι κρίμα που στις 4 Ιουλίου απορρίφθηκε η έκθεση ε, για την, ε, που ήταν σημαντική για την εσωτερική αγορά και τα κοινωνικά θέματα. Ήταν σημαντική ευκαιρία. Πολλά προβλήματα παραμένουν στον τομέα αυτό. Ε, δεν έχουν συντονιστεί οι εθνικοί κανόνε στον τομέα που μα ενδιαφέρει και οι εθνικοί κανόνε δεν εξασφαλίζουν ίσως κανόνε παιχνιδιού για τον τομέα των μεταφορών. Πρέπει όλοι λοιπόν να αποκοινούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να αναζητήσουμε το ίδιο επίπεδο προστασία για τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων. Το καταστημένο που γνωρίζουμε δεν είναι επιλογή. Πρέπει οι εργαζόμενοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι καταναλωτέ να προστατευτούν. Πρέπει να δούμε τώρα τα βασικά ζητήματα, εκεί που απαιτείται συμφωνία. Καμποτάζ, επιστροφή στην ε, χώρα και ούτω καθεξής. Επίσης, Πρέπει να ε, κοιτάξουμε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συγκλίνουν στις απόψεις τους. Εμείς θέλουμε απλώς να διευκολύνουμε εσείς. Η Επιτροπή Τραν ε, μπορείτε να βρείτε συμβαστικέ λύσεις. Μπορείτε να αναζητήσετε το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον με λύσεις για τον ε, το μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κρεμή ζητήματα είναι σαφή. Καμποτάζ, επιστροφή στην χώρα προέλευσης, ανάπαυση στην καμπίνα, στον θάλαμο και άλλα. Θα πρέπει ε, όλοι ε, να ε, κοιτάξετε να επιτύχετε την πρόοδο που απαιτείται για τα θέματα αυτά που υπάρχει ακόμη διαφωνία. Είναι σημαντικό για τους εργαζομένους. Ελπίζουμε ότι η Αυστριακή Προεδρία θα περατώσει τη θέση του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά ώστε να προχωρήσουν και διαπραγματεύσει τον τριμερή διάλογο. Θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη και διαλλακτικότητα στην προσέγγιση και το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για τον ε, τομέα μεταφορών, των οδικών μεταφορών. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας 24 ώρες, 24 ώρα, 7 μέρες τη βδομάδα για να βρεθεί η λύση. Για την ε, κινητικότητα 2. Ε, ευχαριστώ πολύ την κυρία Αγιούτο για την έκθεσή της με τις συνδυασμένες μεταφορές. Ελπίζουμε και σημειώσαμε μάλλον και τη θετική ψηφοφορία στην Επιτροπή Τραν. Ε, η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου ε, ευτυχώς ε, μας εξυπηρέτησε. Αλλά δεν έχουμε ακόμα πετύχει συμφωνία με το πακέτο δικών μεταφορών. Και επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να βρεθεί μια σκόπιμη λύση. Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε και στο Συμβούλιο για να πετύχουμε τον επιδιωκόμενο στόχο. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την απαλλαγή των μεταφορών από τον άνθρακα και ξέρουμε ότι και η Επιτροπή Τραν έχει θετική ε, στάση για το θέμα των καθαρών οχημάτων και έχει πετύχει αρκετά ήδη. Επίσης θέλω να ε, αναφέρω την πρόταση για την αγορά των λεωφορείων και ευχαριστούμε τον κύριο Ζήλα για τη δουλειά του εδώ πέρα. Θα πρέπει όμω να γίνουν αυτή τη στιγμή προσπάθειε και από την πλευρά του Συμβουλίου. Τρίτο πακέτο κινητικότητα. Για να εξοπλιστούμε με τα μέσα, να πετύχουμε ένα σύστημα κινητικότητα που είναι ασφαλέ, καθαρό και αποτελεσματικό για όλου του Ευρωπαίου πολίτε, πρέπει να προχωρήσουμε. Πρώτο κλάδο, η οδική ασφάλεια. Από τι βασικέ προτεραιότητε τη Επιτροπή. Και καταλαβαίνετε γιατί. Παρά τη μεγάλη πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρσι μόνο 25.000 άνθρωποι έχασαν τι ζωέ του στου ευρωπαϊκού δρόμου και ακόμη περισσότεροι τραυματίστηκαν σοβαρά. Τουλάχιστον έξι φορέ παραπάνω. Γνωρίζω ότι η οδική ασφάλεια είναι και για εσά προτεραιότητα και σα ευχαριστώ για την διαρκή σα στεναρή στήριξη. Το πακέτο συμπεριλαμβάνει δύο νομοθετικές προτάσεις που καλύπτουν τις υποδομές και τα οχήματα. Προτείνουμε ένας αριθμός νέων οχημάτων να εξοπλιστούν με τεχνολογία για την ασφάλεια όπως η σωστή λωρίδα, η ευφυής ε, παρακολούθηση της ταχύτητας, ε, το αυτόματο φρενάρισμα και ούτω καθεξής πολλά από αυτά θα εξυπηρετήσουν τους χρήστες των ε, αυτοκινητοδρόμων μας και θα προστατεύσουν και τους πιο ευάλωτους με τα πρόσφατότερα τεχνολογικά επιτεύγματα. Οι κανόνες για την υποδομή της οδικής ασφάλειας και της διαχείρισής της είναι κάτι που πρέπει να ανανεωθεί. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε νέες ε, διαδικασίες γιατί θα πρέπει να δούμε γιατί έχουμε 8% θανάσιμα ατυχήματα και 40% στους βασικούς δρόμους. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και τη χαρτογράφηση όλου του δικτύου. Πρέπει να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια και να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών, ώστε οι διαθεσμικέ διαπραγματεύσει να καταλήξουν σε ένα αίσιο πέρα σύντομα. Για τι δύο ψηφιακέ μα προτάσει, ε, προτείναμε να προχωρήσει και η ε, χρήση των ε, θαλάμων που να βρίσκονται στο μπροστινό μέρος με άθραυστα για μια καλύτερα και για τους οδηγούς αλλά ε, και για του υπόλοιπου χρήστε των αυτοκινητοδρόμων. Για τι ψηφιακέ μα λοιπόν προτάσεις στον τρίτο πακέτο κινητικότητας, για την ενιαία θηρίδα των θαλάσσιων μεταφορών και την ηλεκτρονική ενημέρωση των ε, μεταφορών εμπορευμάτων, θέλουμε να διευκολύνουμε την ψηφιακή διαλειτουργικότητα για τις επιχειρήσεις ε, λογιστική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στιγμή να ξεφύγουμε από το φόρτο και του στήλους από χαρτιά για να περάσουμε σε ηλεκτρονική διαχείριση όλων αυτών και να υπερβούμε τους φραγμούς καθώς και την ε, ζώνη άνεσης όπως τη γνωρίζουν κάποιοι φορείς εδώ στο χώρο. Τέλος, ε, η διαδικασία TNT και η ευθυγράμμισή τους ε, ευτυχώς θα προχωρήσει καθώς μόλις διορίσατε και εσείς οι συζητητές σας. Ευχαριστώ για την ταχεία εξέταση του θέματος σε αυτήν την κοινοβουλευτική θητεία. Γι' αυτό να αναφέρω και μερικά ακόμη κρεμή ζητήματα για την αεροπλοεία. Ξέρω ότι γενικώ έχουμε επιτυχία. Πετύχαμε πρόοδο για τον δίκαιο ανταγωνισμό στο διεθνέ προσκήνιο και ευχαριστώ τον εισηγητή κύριο Τέλιτσκα. Οι τριμερεί διάλογοι έχουν ήδη ξεκινήσει. Η έγκριση του νέου οικονομισμού παραμένει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ύψη τη σημασία να καταλήξουμε σε κανονισμό που να είναι ε, για να έχουμε ένα χρήσιμο εργαλείο σε σχέση με το σημερινό κανονισμό. Ευχαριστώ για τη στήριξή σα ώστε και στο Συμβουλίο να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλο τη χρονιά. Πρόοδο έχει επιτελεστεί και στον τομέα των ε, συμφωνιών για τι μεταφορέ με τρίτε χώρε. Ελπίζω να ολοκληρωθούν κάποιε σύντομα. Η υπογραφή όλων των συμφωνιών έχουν να κάνουν και με το πώ θα ορίσουμε την ευρωπαϊκή επικράτεια. Αυτό απασχολεί πολλέ από τι δημοτεύσει μα και σε αυτό το πλαίσιο να θυμίσω ότι η συνολική και σφαιρική συμφωνία για τι μεταφορέ Ευρωπαϊκή Ένωση Ουκρανία εδώ και πέντε χρόνια δεν έχει εγκριθεί, αλλά αυτό πραγματικά είναι ατυχέ και δεν θα πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Σε ό,τι αφορά την τεχνική, την τεχνική τροποποίηση του κανονισμού 2008-2008 ε, και την, ε, το wet leasing, ε, σημειώνουμε ότι η Επιτροπή Τράν έχει εγκρίνει την έκθεση αυτή, η Αυστριακή Προεδρία έχει ξεκινήσει τι συζητήσει με την ομάδα εργασία άδεια από του 13 Ιουλίου. Οι τριμερεί διάλογοι έχουν ξεκινήσει, θα ξεκινήσουν τον φθινόπωρο. Από τη ρυθμιστική σκοπιά, το ε, θέμα ΣΥΣ 2 ΣΥΝ έχει μπλοκαριστεί στο επίπεδο των ε, διαπραγματεύσεων, των διαθεσμικών διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν κάποιε πτυχέ όμω που δεν θα πρέπει να τι απορρίψουμε, γιατί το σκηνικό τη αεροπλέση έχει αλλάξει. Στηρίζουμε τι προσπάθειε του Κοινοβουλίου με τον ε, βουλευτή κ. Μαρινέσκο για να δούμε πώ μπορεί να προχωρήσει με νέα όθηση ο φάκελο αυτό. Η Αυστριακή Προεδρία θεωρεί μπορεί, θα κοιτάξει μάλλον πότε είναι καλύτερο να οργανώσει συζήτηση για το θέμα αυτό. Ε, ανάλογα με το αποτέλεσμα τη συζήτηση αυτή, η Ρουμανική Προεδρία θα κοιτάξει τι συνέχεια μπορεί να δώσει. Για τα ε, δικαιώματα των επιβατών συνδροδρόμων. Είμαι πολύ χαρούμενο που βλέπω ότι η αναθεώρηση του κανονισμού σα έχει ήδη απασχολήσει και καλωσορίζουμε τι τροπολογίε σα για να αποσαφινιστούν τα δικαιώματα αυτά, ιδίω για την νομική βεβαιότητα και τη σωστή ισορροπία μεταξύ του ρεαλισμού και τη φιλοδοξία που θέλουμε να έχουμε. Βεβαίω, κάποιε από τι τροπολογίε αυτέ αποκλίνουν από του βασικού στόχου που έχουμε θέσει εμεί για του ρυθμιστικού κανόνε από την αναθεώρηση του κανονισμού. Να θυμίσω ότι εμεί θέλαμε μια αναδιατύπωση για να έχουμε μια ταχεία και απλουστευμένη διαδικασία και να πετύχουμε και του στόχου τη καλύτερη νομοθεσία και τη σχετική ατζέντα. Δεν θέλουμε οι διαπραγματεύσει να κρατήσουν πολύ περισσότερο καιρό, γιατί σκοπό είναι να διατυπώσουμε την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών και να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών των δικαιωμάτων και του οικονομικού αντεκτύπου στον τομέα των σιδηροδρόμων η κοινοβουλευτική στήριξη είναι απαραίτητη για να πετύχουμε πραγματικά αποτελέσματα στην κινητικότητα των επιβατών και στην, ε, στην ε, βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων στον τομέα των σιδηροδρόμων. Θέλουμε να υπάρχει ε, βιώσιμη κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική πρόοδος στον τομέα αυτό. Τώρα, η γενική ε, προσέγγιση που εγκρίθηκε στο Συμβούλιο Μεταφορών τον Ιούνιο ε, θα επιτρέψει να επιτελεστεί περαιτέρω πρόοδο όπω και το Κοινοβούλιο έχει καλέσει να γίνει. Ε, για τα θαλάσσια απορρίμματα και λίματα θα πρέπει να κοιτάξουμε να ενισχύσουμε το διεθνέ πλαίσιο με τα απαραίτητα μέτρα. Το ίδιο και για τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Πρέπει να δοθούν κίνητρα και να ενισχυθεί το πλαίσιο που ελέγχει το σύστημα διαχείρισης και αποκομιδής των αποβλήτων. Η κυρία Μάισνερ μα βοήθησε πολύ στο θέμα αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει ότι η έκθεση αυτή θα εγκριθεί σύντομα για να ξεκινήσουν και τριμερείς διάλογοι και να προχωρήσει τελική συμφωνία μέχρι την επόμενη χρονιά. Και δύο κουβέντες για το Brexit, διότι όπως ξέρετε είναι και περίπλοκο και λεπτό το ζήτημα. Το Brexit μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις μεταφορές, κυρίως εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη, του και το γενικό κοινό για του αντικτύπους μπορεί να έχει το Brexit στου διάφορου τρόπου μεταφορών. Τα διάφορα, οι διάφορε συνέπειε που μπορούν να προκύψουν από το ε, Brexit είναι ζωτική σημασία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις εθνικές, στα εθνικά κράτη και στο επίπεδο των ενδιαφερομένων για να αποκριθούμε στι νέε προκλήσει. Δύο νομοθετικέ προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπό έχουν να ε, καλύψουν τι ανάγκε του βασικού δικτύου διαδρόμων του TNT και των θαλάσσιων μεταφορών τα κοιτάζουν και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα προτινόμενα μέτρα. Ελπίζουμε να προχωρήσουμε με, με πήγοντα τουλάχιστον μέτρα τι ερχόμενε εβδομάδε για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλε τι υποθέσει Brexit τι ερχόμενε εβδομάδε. Ε, εν είδε συμπεράσματο, Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτέ, ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη διαρκή σα στήριξη τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Καθώ πλησιάζουμε στο τέλο τη θητεία και του Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να αναγνωρίσουμε την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε μεταξύ τη Επιτροπή Τραν και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερο από ποτέ πρέπει να διατηρήσουμε αμύωτα αυτό το ρυθμό και τη στενή μα συνεργασία του τελευταίου αυτού μήνε σε τόσο ζωτικά ζητήματα όπω την χρηματοδότηση των μεταφορών και τα πακέτα κινητικότητα. Πραγματικά αναμένω διακαώ τι ερωτήσει και τα σχόλιά σα και θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω στο χρόνο που μα απομένει. Τα σημείωσαν και οι συνάδελφοι από εδώ δεξιά και αριστερά και πρόεδρε ε, παρακαλώ αν θέλετε συγκεκριμένα απάντηση από μένα μπορείτε να μου το ζητάτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρουλάη για αυτή την, ε, αυτό το άπλωμα του θεματολογίου για το επόμενο οκτάμινο. Και καλώς ορίζω τους ε, προσκεκλημένους του φίλου Ντομίνη Τρικέ 18 επισκέπτες από την SNCF, τους γαλλικούς σιδηροδρόμους στην αίθουσα. Σηκωθείτε να σας δούμε και να σας καλωσορίσουμε. Ε, την πατήσατε. Νομίζατε ότι θα μπείτε και θα βγείτε διακριτικά από την αίθουσα, αλλά όχι. Κύριε Λολάη, Πριν περάσουμε στη συζήτηση για τα θέματα αυτά, θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο φέτος κατά κάποιο τρόπο με παρηγόρησε κιόλα μετά την κατάρρευση της γέφυρας στην Γένοβα, αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Ένας υπουργό της Ιταλίας βγήκε και είπε «Πταίει η Ευρώπη» και ευχαριστώ την Επιτροπή που βάζει τα πράγματα στη θέση του, τους. Γιατί αυτή η τραγωδία δεν οφείλεται στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια πολιτική επιλογή που δεν ελήφθη. Δηλαδή δεν ελήφθη απόφαση να μπουν ως προτεραιότητα τα τελευταία 10 και 20 χρόνια, όχι φέτος, οι υποδομές, οι οδικές, οι γέφυρες, επενδύσεις που χρειάζονται για την ασφάλεια των συμπολιτών μας, δεν είναι δυνατόν να λέμε δεν γίνανε επειδή φταίει η Ευρώπη. Και ευχαριστώ την Επιτροπή μόνο τώρα έτσι μην το πάρετε και επάνω σας, που αντιδρά εγκαίρως, διότι αν αφήνουμε να περνάει ο καιρός και να δίνεται η εντύπωση ότι φταίει η Ευρώπη, δεν προχωράει το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και κάτι ακόμα να γίνονται τόσα και τόσα, έγιναν αυτό το καλοκαίρι ιδιαίτερα, όσο λείπαμε. Ένα άλλο λοιπόν, αυτή η διαβούλευση με τους πολίτες για την οποία θέλω να σας ευχαριστήσω, για την αλλαγή της ώρας επιτυχία μεγαλειώδης. Η μεγαλύτερη εκδήλωση ε, διαβούλευσης με τους πολίτες στην Ευρώπη. 4,6 εκατομμύρια πολιτών μέσα σε δυο 3 ε, εβδομάδες ανταποκρίθηκαν. Και ο κύριος Γιούγκερ, να, είπε, πολύ καλά, ακούμε αυτά που έχουν να μας πούν οι πολίτες. Και καλά κάνει η Ευρώπη με τις διαβουλεύσεις αυτές, τα ευρωπαϊκές εργαλεία τα οποία βοηθούν και τη δική μας τη δουλειά και παρακολουθούν και συνοδεύουν τη δική μας τη δουλειά εδώ της Επιτροπής των Μεταφορών. Σας ευχαριστώ λοιπόν και για αυτή την πρωτοβουλία. Ξεκινούμε τη συζήτηση. Με πρώτο πρώτο τον κύριο Φαντενκάμπ που έχει μόνο τρία λεπτά στη διάθεσή του, αλλά ξέρω πόσο λακωνικός μπορείτε να είστε, κύριε Φαντανκάμπ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ρωτώ με. Μήπως θα έπρεπε να σταματήσουμε τη συνεδρίαση και να ανοίξουμε καμιά σαμπάνια. Με αυτά που μας λέει ο κύριος Ρολάι. είμαστε πραγματικά στο ζενήθ. Είμαστε η, κατα... καταπληκτικότερη επιτροπή του κόσμου. Για τις μεταφορές αλλάζουν με τα πάντα προς το καλύτερο. Ε, είπατε και εσείς ότι, είμαστε, ε, ότι έχουμε την τάση να αντιδρούμε στα προβλήματα, όχι να τα προλαβαίνουμε. Πρέπει όμως και να προσέχουμε εμεί τον κοσμάκο το δικό μας το μικρό που ζούμε να μην ε, ε, επενούμε τόσο πολύ αυτούς, να μην αυτοσυγχαιρόμαστε, γιατί δεν είναι ακριβώς τα πράγματα όπως μας τα λέει ο κύριος Σορολάη. Στην παρέμβασή του πολλές φορές ε, απευθύνθηκε προς το Συμβούλιο. Ξέρουμε ότι, στην, ότι μεταξύ μας Επιτροπή και Κοινοβούλιο συχνά συμφωνούμε και έρχονται τα κρατη να παρεμποδίσουν ε, κάποιες εργασίες και την πρόοδο ε, που εμείς θέλουμε να προωθήσουμε. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Έχω κάποιες ερωτήσεις λοιπόν και χωρίς να θέλω να ταράξω τα νερά της ευτυχίας, έχουμε τα πακέτα κινητικότητας 2 και 3. Έχουν περάσει έξι μήνες. Είχαμε κάποια χρόνια για να επεξεργαστούμε τα θέματα αυτά, των πακέτων 2 και 3. Αφήσαμε να περάσει όμως ο καιρός και ενώ θα πούσουμε να τα έχουμε προχωρήσει πολύ νωρίτερα, έρχεται τώρα η ώρα. Κοινωνικό ταμείο. Όλο και μικρότερη η χρηματοδότησή του. Σε όρου προπολογισμού. μιλούμε για τρέχουσες τιμέ, για σταθερέ τιμέ κτλ. Για το MIE που ωστόσο είναι μια από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις, από τα πιο επιτυχημένα εγχειρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Επίσης βιωσιμότητα και μεταφορές. Είστε ειδικό από ό,τι ξέρω, ειδικά των ε, αεροπορικών μεταφορών. Η ΚΑΟ λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς ε, πρόκειται να συνεργαστούν στον χώρο των μεταφορών για να περιορίσουν τις εκπομπές πάνω απ' όλα. Οι θαλάσσιες μεταφορές επίσης που επίσης έχουν πολύ επιβαρυντικές εκπομπές. Και ξαναγυρνώ στο πακέτο κινητικότητας υπαριθμών 1. Το συζήτησαμε πολύ στις ε, συνεδριάσεις των συντονιστών μας. Όλοι αρχίζουν λοιπόν και εξοπλίζονται από ό,τι βλέπουμε, όλοι αρχίζουν και ετοιμάζονται για να ανασκουμποθούμε και να αντιμετωπίσουμε το πακέτο για την κινητικότητα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το κλείσουμε. Το Νοέμβριο στην Ολομέλεια ελπίζουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι για να ψηφίσουμε. Βεβαίως πρέπει να υδρώσουμε για να τα καταφέρουμε. Έχουμε πολλή δουλειά, αλλά ελπίζω να μην εγκαταλείψετε το φάκελο αυτό σε αυτή τη χρονική στιγμή, κύριε Ρολάη, και ό,τι επένδυση έχει γίνει σε ενεργητικότητα και δουλειά να αξιοποιηθεί. Ευχαριστώ, κύριε Φαντενκάμπ, και πάνω απ' όλα που σεβαστήκα το χρόνο. Κύριε Αρτού, τρία λεπτά επίση. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ ήρθατε, κύριε Ρολάη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα είπατε. Έχω τρει ερωτήσει και ε, σα τι παρουσιάζω ευθύ αμέσω. Πρώτα απ' όλα ένα θέμα πολύ σημαντικό για μένα, για όλους μας, οι υποδομές που σχεδιάζουμε για το μέλλον και κυρίως ή με, με χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Ε, CLG, LNG, υδρογόνο, ηλεκτρικό, όλα αυτά λοιπόν που θα μας επιτρέψουν και να υλοποιήσουμε τους στόχους της ε, ε, εκμυδένισης των εκπομπών άνθρακα. Το έχετε εσείς ως Επιτροπή μελετήσει και προωθήσει. Πολύ καλά βήματα, 800 εκατομμύρια βλέπω και είμαστε ευγνώμονες μεν, ωστόσο είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν αρκούν. Με τους και ηγητές λοιπόν και επί τη ευκαιρία της έκθεσης πρωτοβουλίας που έχω αναλάβει, συζητήσαμε το πώς μπορούμε να δώσουμε περισσότερη όθηση, πώς μπορούμε να απαιτήσουμε 2,5 συνολικά δισεκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο προϋπολογισμό που θεωρούμε δυνατόν να εξασφαλιστούν ε, γιατί τελικά θα πρέπει βέβαια ο ιδιωτικό τομέα να αναλάβει το μερίδιο του λέοντο τη χρηματοδότηση. Μπορείτε λοιπόν εσεί να δείτε κάποιε λύσει καταρχά ω προ τη χρηματοδότηση και την προώθηση αυτών των έργων υποδομών. Και επίση ο Επίτροπο Γιουνκέρ έχει εκδηλώσει τη, βούληση, τη βούληση να ε, ζητήσει τη γνώμη των ε, πολιτών, των 500 εκείνων χιλιάδων που έχουν συμμετάσχει στην διαβούλευση και πολλών άλλων που δεν περίμενα εγώ να ε, ανταποκριθούν. Η διαβούλευση λοιπόν αποδεικνύεται ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και πρέπει να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, επόμενες εβδομάδες. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, μπορούμε να περιμένουμε μια νομοθετική πρόταση για το θέμα αυτό. Και στις αεροπορικές μεταφορές τελευταίο σημείο, γιατί η Επίτροπος Μπούρτς μας είχε μιλήσει για την εισαγωγή συμπερίληψη της κοινωνικής διάστασης στις αεροπορικές μεταφορές. Μία πρόταση που είχε ξεκινήσει με τη στρατηγική για τις αερίες μεταφορές το 2015, που όμως εντωμεταξύ δεν είδαμε τίποτε συγκεκριμένο να παρουσιάζεται ως πρόταση. Υπάρχει μία μελέτη που έχετε εσείς ως Επιτροπή αναθέσει, η οποία ιδιαίτερα στέκεται στις ατυπικές μορφές εργασίας, στις ε, συμβάσεις μηδενικών ορών, της, ε, την ανατροπή των ε, εργασιακών σχέσεων που μάλιστα χαρακτηρίζει ως την κορυφή του παγόβουνου και ρωτώ εσείς κύριε λέει τι ιδιαίτερη έμφαση μπορείτε να θέσετε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κοινωνική διάσταση και το κοινωνικό ντάμπινγκ που βλέπουμε να πραγματοποιείται στις αεροπορικές μεταφορές. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φώστορ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ κύριε Λουλά, ήταν πολύ πλήρης η ε, ενημέρωση που μας προσφέρατε. Προφανώς είναι πολλά τα θετικά, τα επιτεύγματα. Υπάρχουν όμως ακόμη τομείς που χρειάζονται περισσότερη επεξεργασία το πακέτ, τα πακέτα κινητικότητας, αλλά βέβαια πιστεύω ότι όπου, όποιος θέλει μπορεί. Έτσι λοιπόν, ε, στο επόμενο διάστημα έχουμε να καταγράψουμε πολλά θετικά. Εγώ προσωπικώς είμαι υπερήφανη για τα όσα έχουμε επιτύχει στις μεταφορές ε, και με την Επιτροπή φυσικά, χωρίς πάντα να είμαστε σύμφωνοι, αλλά τα καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ε, συμφωνώ με τα σχόλια του Wim van den Kamp στο θέμα με το κοινωνικό ταμείο. Και βέβαια ε, πολίτε στην δημοσιονομικό πλαίσιο, Ταμείο Συνοχής ε, και γενικά οι προοπτικές που βλέπουμε μας αποδεικνύουν ότι πρέπει εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών να απαιτήσουμε να έχουμε για όλα τα μεγάλα έργα τις απαραίτητες, ε, τους απαραίτητους σπόρους, γιατί είναι προς το συμφέρον όλων. Με καλές υποδομές μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους στόχους και τους περιβαλλοντικούς και των μεταφορών της κινητικότητας τα λοιπά. Έχουμε πολλά προβλήματα και ρήπανσης ε, του ατμοσφαιρικού αέρα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε χάρη σε καλέ υποδομέ. και θα, γνωρίσω, θα γυρίσω στο αγαπημένο μου θέμα που γνωρίζετε πολύ καλά ποιο είναι, το χώρο των εναέριων μεταφορών. Πολύ σωστά λέτε ότι η Άσα έχει προχωρήσει σε μια ε, αναθεώρηση που πρέπει και εμείς ε, να προωθήσουμε, η ΕΑΣΑ μάλλον έχει προχωρήσει την αναθεώρηση, πρέπει και εμείς να προωθήσουμε, ε, δεν πρέπει να καθυστερήσουμε περισσότερο. Αλλά με ανησυχεί ιδιαίτερο το γεγονός ότι ο κανονισμός 261 έχει παραμείνει ανενεργός και μπορούμε να πούμε βεβαίως ότι το Συμβούλιο δεν έχει την πολιτική βούληση να προωθήσει τα θέματα του κανονισμού αυτού. Από την άλλη βέβαια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε, διατύπωσε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα επέτρεπαν να προχωρήσουν τα θέματα αυτά. Αλλά ξέρουμε ότι νομικά ε, αυτό σημαίνει πως έχουν μείνει ζητήματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί στα κράτη-μέλη ή που αντιμετωπίζονται κατά πολύ κατακαιρματισμένο τρόπο και βέβαια όλη αυτή η κατάσταση είναι ε, ένα συνονθήλευμα προβλημάτων. Επίσης, έχουμε μια σειρά από απροειδοποιητές απεργίες ε, στα κράτη-μέλη, στις ενέργειες μεταφορές. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα κράτος μέλος, αλλά ξέρουμε πιανού η συμπεριφορά είναι αυτή η οποία οδηγεί στην ε, ε, εβδομαδιαία ανάδειξη απροειδοποιητών απεργιών στι εναέριε μεταφορές τελευταία στη Γαλλία και εν πάση περιπτώσει δεν έχουν γίνει συλλογικέ διαπραγματεύσει. Και βεβαίω δεν πρέπει να λησμονούμε ότι μπορεί να έχουμε δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και των καταναλωτών δικαιώματα υπάρχουν και τέτοιου είδους ε, διαταραχή των ε, ε, μεταφορών εις βάρος του καταναλωτή είναι απαράδεκτη. Πρέπει λοιπόν να εκδηλωθεί η πολιτική βούληση και να εξευρεθεί ο δρόμος ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα. Ξέρουμε ότι κάποια κρατή-μέλη έχουν τελικά την ε, ευθύνη της εξασφάλισης των υποδομών. Χρειαζόμαστε περισσότερους διαδρόμους, ε, προσγείωσης απογείωσης, περισσότερες υποδομές γενικά και τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσουν και πρέπει να το καταφέρουν καλύτερα από ό,τι μέχρι τώρα. Και επιπλέον, Πρόεδρε, για να συνεχίσω, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριο Ολολάη, και ευχαριστώ ε, και ελπίζω ότι τα θέματα αυτά θα, θα ε, αντιμετωπιστούν μέχρι το τέλος ε, της εντολής μας. Ευχαριστώ τα για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Καταρχήν, Εκτιμώ ιδιαίτερα την πλήρη επισκόπηση που μας έκανε ο Γενικός Διευθυντής της ΜΟΥΒ και να συμφωνήσω με τα περισσότερα σχόλιά του. Μίλησε για το πολιτικό προφίλ των μεταφορών, πόσο σημαντική είναι η εικόνα για τις μεταφορές. Και είχαμε και τις ημέρες των Διευρωπαϊκών Δίκτυων Μεταφορών, έτσι προωθούμε τις μεταφορές και τις προβάλλουμε όσο γίνεται. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία στην θετική αυτή προβολή των μεταφορών. Ε, και σίγουρα θα πρέπει να περάσει το μήνυμα για τις βελτίσεις των μεταφορών και στο κοινό. Οι συντονιστές των TNT όταν μας μιλούν ή εδώ ή αλλού δεν καταλαβαίνουμε πόση πρόοδο έχουμε σημειώσει. Φανταστείτε, δεν καταλαβαίνουμε εμείς πώς είναι δυνατόν να αντιληφθεί το κοινό την πρόοδο. Μιλούμε για καταμέτρηση, για δείκτες, για παρακολούθηση, για επικοινωνία καλή. Πρέπει να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας με τους Ευρωπαίους πολίτες και να προσέχουμε τη διατύπωση χρησιμοποιούμε ε, στην επικοινωνία μας με το κοινό. Γιατί μερικές φορές ε, ο τρόπος που προωθούμε ή προβάλλουμε κάτι να μην ε, μας θυμίζει την προπαγάνδα πριν το 89. Προσοχή λοιπόν, μία ευαισθησία στον τρόπο που επικοινωνούμε με το κοινό αυτό που μας προβληματίζουν μερικές φορές είναι τα επίπεδα χρηματοδότησης και θα πρέπει και εκεί να βελτιωθούμε. Και περιμένω ε, την ομιλία του ε, Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση της Ένωσης. Ελπίζω να κατάλαβε επιτέλους τη σημασία που έχουν οι μεταφορές στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήθελα καλύτερη προβολή και περισσότερη υποστήριξη των μεταφορών, γιατί πρόκειται για ένα κλάδο που είχε μεγάλη επιτυχία και επηρεάζει την ανάπτυξη, την καθημερινότητα των πολιτών, τις επιχειρήσεις, οπότε ελπίζω να έλαβε το μήνυμα ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να φανεί αυτό στην επόμενη το μιλή για την κατάσταση της Ένωσης. Σε ό,τι αφορά το πακέτο κινητικότητας, φυσικά θέλουμε να προσφέρουμε έργο και σίγουρα στις 4 Ιουλίου χάσαμε μια ευκαιρία. Α, θέλουμε πρόοδο, αλλά όχι πάση θυσία. Και πρέπει η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιληφθεί ότι προτιμούμε να μην έχουμε νομοθεσία παρά κακή νομοθεσία. Δεν θέλουμε ε, μονομερή μέτρα των κρατών μελών που θα είναι εις βάρος κοινή αγορά. αλλά θέλουμε ισορροπημένο αποτέλεσμα. Αναφέρθηκε ο κανονισμός 868, δεν μπορώ να επισέλθω τώρα σε πολλές λεπτομέρειες, ελπίζω να τα καταφέρουμε και τρία σύντομα σχόλια στο τέλος. Καταρχήν θα εκτιμούσε ιδιαίτερο αν προς το τέλος της ΕΤΕΣ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήσει μια παρακαταθήκη για το μέλλον για να μας πει πού θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, να αφήσει ένα πολιτικό έγγραφο με την πολιτική της παρακαταθήκη και κάτι που θα είναι με την πολιτικη της παρακαταθηκη και κατι που θα ειναι βαναγνωστο για να καταλάβει και ο κόσμος πού σημειώσαμε πρόοδο, πού θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για να μην χάσουμε και άλλη ευκαιρία. Και χαίρομαι επίσης για τη στρατηγική για την αεροπορία. και αυτό αναφέρεται σε πολλά πολιτικά έγγραφα. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά το δίκτυο κινητικότητας. Σημειώσαμε πρόοδο, το είπαμε και στο Τάλιν. Φαίνεται ίσονο σημασία, αλλά είναι πολύ σημαντικό θέμα για κάθε μηχανισμό της πολιτικής μεταφορών. Θα πρέπει να το ενημερώσουμε αυτό το δίκτυ. Σε ό,τι αφορά το Brexit, ε, το ξέρω ότι έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες και ο Μισελ Μπαρνιέ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικώ και στις διάφορες ομάδες εργασίας ε, θα ήθελα να ε, είναι σαφές και στην νομοθεσία τι μας περιμένει. Χωρίς να παρέμβουμε στη διαπραγμάτευση γιατί για τον Brexit θα πρέπει να ενημερωθούμε για τον αντίκτυπο θα έχει στα επιμέρους νομοθετικά πακέτα. Σε ευχαριστούμε κύριε Τελίσκα. Ε, έχετε ξεπεράσει το τρίλεπτο, αλλά βλέπουμε από τον τρόπο που μιλάτε τι πάθος ε, σας διακατέχει για τα θέματα αυτά. Γι' αυτό σας επέτρεψα να υπερβείτε λίγο το χρόνο σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και τον ε, Γενικό Διευθυντή της ε, ΜΟΥΒ για την προθυμία του να μας μιλήσει και να απαντήσει στις απορίες μας. Ε, πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τις ενέργειες μεταφορές αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση και στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Το τρένο είναι φθηνότερο, γιατί να μην το προωθήσουμε. Βέβαια τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να κλείσει κανείς ε, εισιτήριο αεροπορικό παρά σιδηροδρομικό. Θα πρέπει λοιπόν να ε, βοηθήσουμε ε, την κατάσταση, να διευκολύνουμε την, τις κρατήσεις και στις σιδηροδρομικές μεταφορές γιατί πολλές φορές όταν έχουμε και διασυνοριακά ταξίδια, ε, θα πρέπει να βγάζουμε τα επιμέρους εισιτήρια ξεχωριστά στην κάθε χώρα. Ε, και κάτι τέτοιο είναι πολύ χρονοβόρο, ενώ στις αεροπορικές μεταφορές είναι πολύ πιο εύκολες οι κρατήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε τις κρατήσεις τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διασυνοριακά ταξίδια. Πιστεύω ότι αν βελτιώσουμε το σύστημα κρατήσεων στους σιδηροδρόμους, θα ενθαρρύνουμε τους πολίτες ε, να προσφεύγουν περισσότερο στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Γιατί πολλές φορές ε, οι σιδηρόδρομοι είναι μονοπόλια και κάπως κλειστά στη συνεργασία. Θα πρέπει αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Επίσης θα πρέπει οι σιδηροδρομικές εταιρείε να ανοίξουν τα δεδομένα τους και να είναι πιο ανοιχτές στη συνεργασία. Έτσι όλοι θα εποφεληθούμε από πρόθεση των σιδηροδρομικών μεταφορών και θα πρέπει να έχουμε αντίστοιχε τιμές ή ε, να είναι εύκολη σύγκριση των τιμών από το χρήστη. Γιατί να έχουμε τέτοια διαφορετική μεταχείριση στο σιδηροδρόμο σε σχέση με τι ενέργειε μεταφορέ. Ελπίζω να αναλάβει σχετικέ πρωτοβουλίε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κύριε Νταλούντε. Η ε, κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ το Διευθυντή που είναι εδώ. Τα κύρια σημεία, λοιπόν. Πρώτον, για το Κοινωνικό Ταμείο και τους... Για το συνδέοντα στην Ευρώπη και τους πόρους για την ε, Νότια Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως, αλλά εγώ αναφέρομαι σε όρους ασφάλειας για τους πολίτες Ευρώπης μπορεί να μην ε, αρκούν οι πόροι όταν ε, ε, το συνδέοντας Ευρώπη στηρίζεται περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα, στον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφορών πορών και έτσι υπάρχουν κάποια σημεία του κεντρικού δικτύου που ευνοούνται σε σχέση με άλλα. Γιατί οι αποφάσεις λαμβάνονται από, την, από τις Βρυξέλλες και για το τρένο υψηλή ταχύτητα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Ερωτώ λοιπόν, αυτό ο κίνδυνο δεν υπάρχει και στην προσεχή, στον προσεχή προγραμματισμό, δηλαδή να ευνοηθεί περισσότερο το κέντρο και οι ανατολικέ χώρε Ευρώπη και να αποκλειστούν από το σχεδιασμό ε, οι υποβαθμισμένε περιοχέ και κυρίω ο νότο Ευρώπη. Ξέρω βεβαίω ότι πρέπει να γίνονται και εθνικέ επιλογέ, αλλά ε, η Ιταλία μένει μόνη τη στη χρηματοδότηση των ε, δικτύων στον Νότο. Ενιαίοι εθέρες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχει ολοκληρωθεί κανένας από τους τέσσερις κύριους στόχους. Τα στοιχεία δεδομένα, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα σημαίνουν οικονομία κλίμακας, όλο και περισσότερο, κριτήρια οικονομικά δηλαδή. Και έτσι κλείνουν κέντρα ελέγχου στην Πάντοβα, στο Πρίντιζι, που μετατρέπονται σε απομακρυσμένους πύργους ελέγχου. Ρωτώ λοιπόν, δεν πρέπει ο ενιαίος ουρανός, ο ενιαίοι θέρες τουλάχιστον να περάσουν μέσα από έναν επανέλεγχο πριν την προώθηση νέων προγραμμάτων και σχεδίων. Δεν πρέπει να επαληθευτεί μη τυχόν και προκύπτουν κίνδυνοι για την ασφάλεια όταν έρχεται η ώρα της υλοποίησης, ε, της εκκίνησης μάλλον της προσεχούς ε, περίοδου αναφοράς, της νούμερο 3, για το προσωπικό, για το πλήρωμα και τις ατοπικές ε, μορφές απασχόλησης στους εργαζομένους σε αέριες μεταφορές. Έχει γίνει τίποτα και άλλα 30 δευτερόλεπτα για την κινητικότητα όταν προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα στις οδικές μεταφορές, πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε το καμποτάζ, την, ε, το κοινωνικό ντάμπινγκ, συνθήκες δουλείας υπό τις οποίες αναγκάζονται να εργάζονται οι οδηγοί στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να υπάρξει μια λύση που για μας θα έπρεπε να είναι η λύση που έχει προτείνει η Επιτροπή Απασχόλησης. Έλεγχη, αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη, χρήση της τεχνολογίας Ταχογράφη και GNSS. Το Κοινοβούλιο του Σέλος θα πρέπει να ξεπεράσει τις ε, κομματικές ε, και προεκλογικές, ε, τους προεκλογικούς διχασμούς και να βρει μια ενιαία θέση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάτο για την παρέμβασή σας και επανέρχομαι στον κύριο Ρουλάη που θα μας απαντήσει. Παρακαλώ. Ήταν πληθώρα τα σχόλια των συντονιστών μας, έτσι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά τους συντονιστές για τα σχόλιά τους και τις ερωτήσεις τους. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Πρώτα όμως θα ήθελα να ξεκινήσω με τα δικά σας σχόλια και να σε ευχαριστήσω για τα ευγενικά σας λόγια Είδατε όντως ότι ε, το καλοκαίρι η κατάρρευση της ε, γέφυρας στη Τζένοβα ήταν πραγματικά τραγωδία και ήταν πολλές οι ε, συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την ε, τραγωδία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν τμήμα του προβλήματος, είναι όπως συνήθω με τις λύσεις. Και χαίρομαι για τον τρόπο που διατυπώσατε το σχόλιο σας για το θέμα αυτό. Επίση, ευχαριστώ για το σχόλιο σα για τη θερινή ώρα. όντω. ήταν μια προηγούμενη εμπειρία, πρωτοφανή. Θα θυμάστε ότι όταν ξεκινήσαμε τι διαβουλευσει, ήδη από τι πρώτε μέρε είχαμε πρόβλημα λόγω της συμφόρησης ε, στα συστήματα πληροφοριών. Δεν φανταζόμασταν να έχουμε τόσες ε, να κατακλειστούμε από τόσες ε, πληροφορίες. Είχαμε πάνω από 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις και πραγματικά ήταν πολλαπλάσια η η αντίδραση του κοινού. Ήταν τεράστιο το ενδιαφέρον ε, των ε, Ευρωπαίων πολιτών για το θέμα αυτό και σκεφτήκαμε πώς θα τους αναμίξουμε, πώς θα τους δώσουμε την ευκαιρία να επηρεάσουν την πολιτική μας και να μπορέσουν να δουν και εκ των υστέρων την έκβαση. Ε, ευτυχώς διορθώσαμε πολύ γρήγορα τα προβλήματα πληροφορικής λόγω της συμφόρησης που παρατηρήθηκε στα δίκτυα και έτσι μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τη διαβούλευση. Επίσης, προλάβατε κάπως την απάντηση που θα έδινα στον κύριο Αρτούκ, γιατί και εκείνο ρώτησε για τη θερινή ώρα και τι θα κάνουμε με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων. Νομίζω ότι κατέστησα φες ότι και η Επίτροπος Μπούλτς και ο Πρόεδρος Γιούνκερ ε, δήλωσαν ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μας και συζητήθηκε και στο σεμινάριο τη ευρωπαϊκή επιτροπή Επιτροπής. Εκεί ο πρόεδρο είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεωρήσει τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Αυτό εξετάζει τώρα και ολοκληρώνει την ανάλυση των διαβουλεύσεων που θα δημοσιεύσει τις επόμενες εβδομάδες. Του τέστην, άμα ρωτάτε αν θα ισχύσει η διαδικασία συναμόφασης, λέω ναι, θα υποβάλουμε πρόταση και κατά πάσα πιθανότητα η πρόταση θα λάβει υπόψη απόψη των Ευρωπαίων πολιτών και την έντονη προτίμησή τους υπέρ της κατάργησης ε, της αλλαγής της ώρας. Και ταυτόχρονα με το πνεύμα της επικουρικότητας και αφήνουμε τα μικρά στην τοπική κλίμακα και στα κράτη-μέλη ε, θα αποφασίσουμε ποια ώρα θα καταργήσουμε και ποια ώρα θα κρατήσουμε. Πάντως η απάντησή μου είναι ότι βεβαίως θα υποβάλουμε πρόταση ε, μετά την δημοσίευση της ανάλυσης ε, των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης. Και γιατί επιταχύναμε τη διαδικασία, γιατί θέλαμε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει την ευκαιρία να αποφανθεί. Γιατί αν το αφήναμε να καθυστερήσει, δεν θα προλάβαινε το Ρινό κοινοβούλιο να αποφανθεί. Οπότε εσείς θα αποφασίσετε ε, ποια θα είναι τελική έκβαση για τους Ευρωπαίους πολίτες ως προς την ώρα. Κύριε Λαλέη, μία μικρή διόρθωση. Αν μπήκε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη αλλαγή της ώρας, αυτό έγινε χάρη στην Επιτροπή Μεταφορών. Εμείς εκπονήσαμε και εγκρίναμε το σχετικό ψήφισμα, οπότε ε, ε, είπατε ότι θα πρέπει εμεί να αποφανθούμε, αλλά αυτό έγινε χάρη σε εμά που πήραμε την πρωτοβουλία με το ψήφισμά μα. Όλα από εμά ξεκίνησαν και φυσικά προχωρούμε σε συνεργασία και συμβαδίζουμε. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά με αποθάρρυνε πριν ο κύριος Βαντερκάμ είπα να μην είμαι τόσο θετικός για το έργο της Επιτροπής, γι' αυτό δεν σας ανέφερα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά όντω η Επιτροπή σα έπαιξε κέριο ρόλο και εσείς προωθήσατε τη, ουσιαστικά και εθαρρύνετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περάσει στη διαβούλευση. Τώρα, κύριε Βάντερ πιστεύω ότι θα πρέπει να μην μιλάμε μόνο για τα κενά και τις αποτυχίες μας, αλλά να προβάλλουμε και τις επιτυχίες μας και τα επιτεύγματά μας. Και όντως είμαστε αρκετά μετριόφρονες εδώ ε, θα πρέπει να επικοινωνούμε καλύτερα την πρόοδο και τα πλεονεκτήματά μας. Εγώ είμαι εκφύσεως αισιόδοξο άνθρωπος και βλέπω πάντα το ποτήρι μισογεμάτο και βλέπω τα επιτεύγματα και θα πρέπει να τα αναδεικνύουμε και να το υπενθυμίζουμε. Και πιστεύω ότι ήταν θετικό το πρόγραμμά μας και θα συνεχίσουμε να το εφαρμόζουμε σε συνεργασία μαζί σας και κυρίως σε συνεργασία με την Επιτροπή Μεταφορών. Επίσης, μιλήσατε για τα για το δεύτερο και τρίτο πακέτο κινητικότητα και αν μπορούσαμε να είχαμε επιταχύνει του ρυθμού. Ναι, θα μπορούσαμε, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε την ποιότητα, την ανάγκη του ευνομοθετήν και να λάβουμε υπόψη και τι διαδικασίε που μερικέ φορέ είναι χρονοβόρε. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ένα ισορροπημένο πακέτο ποιοτικό και ουσιαστικό. Και πάντα γίνεται μια κούρσα. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της ταχύτητας και της ποιότητα. Όποιο βιάζεται αυτή μερικέ φορέ. Δεν θα πρέπει να θυσιάζουμε την ποιότητα στο βωμό τη ταχύτητα. Φυσικά πάντα μπορούμε να είμαστε καλύτεροι και ταχύτεροι, αλλά τα πράγματα έχουν όσα έχουν και σίγουρα η πρόταση θα μπορούσε να είχε οριμάσει λίγο περισσότερο, αλλά νομίζω ότι χρειάστηκε αυτό ο χρόνο όριμα για να έχουμε και καλή ποιότητα, καλό αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά το συνδέοντο στην Ευρώπη, ήταν πολύ καλό αυτό το εργαλείο. Πολύ καλή αυτή η διευκόλυνση και εσείς ε, συμμετείχατε στα σημαντική συνιστόσα του ιδέατος στην Ευρώπη και συμμετείχατε σε διάφορες εκδηλώσεις και σε συζητήσεις που έγιναν για το μέλλον του συνδέοντος στην Ευρώπη. Συμβάλλατε τα μάλα λοιπόν ε, και ε, είστε κι εσείς ε, υπεύθυνοι για αυτή την καλή πρόταση. Φυσικά ο προπολογισμό θα μπορούσε να ήταν πιο μεγάλος. Πάντα υπάρχει δυνατότητα για ε, μεγαλύτερο προπολογισμό, αλλά τουλάχιστον κρατήσαμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και συνολικά στον προπολογισμό έχουμε λιγότερα κονδύλια, οπότε πρέπει να κάνουμε κάποιες επιλογές. Και Όπω ξέρετε, περικοπές έγιναν στι περισσότερες δημοσιονομικές γραμμές, ενώ στο ιδιαίτερα στην Ευρώπη δεν έγιναν περικοπές. Μπορεί να μην έχουμε αύξηση του προπολογισμού, αλλά τουλάχιστον δεν είχαμε μείωση του προπολογισμού όπως έγινε σε άλλες πολιτικές. Και ούτως ή άλλως δεν έχει τελειώσει η συζήτηση για το συνδέοντα στην Ευρώπη συνεχίζεται και οι διαπραγματεύσει, συνεχίζονται και το Συμβούλιο θα πρέπει από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίζουν για την τελική έκβαση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Και φαντάζομαι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίζει ε, να στηρίζει την ανάγκη φιλόδοξου προπολογισμού για το σύνθετο στην Ευρώπη, για τις απαραίτητες επενδύσει. Και μάλιστα είπα 350 δι μόνο για το βασικό δίκτυο. Και φυσικά θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα για τι μεταφορέ, αναμφίβολα, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε και άλλες ε, νέες προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετανάστευση, προστασία ε, των ε, εργαζομένων και ούτω καθεξής. Οπότε θα πρέπει να προβλέψουμε κονδύλια και για αυτές τις προκλήσεις. Να βρούμε τη σωστή ισορροπία λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα η Επιτροπή σας θέτει τις μεταφορές στη, ως προτεραιότητα του θεματολογίου και του προγράμματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και το θέμα της βιωσιμότητας των μεταφορών είναι πολύ σημαντικό και βρίσκεται στο επίκεντρο και του δικού μας έργου και προβληματισμού και η Επίτροπος Μπούλτς ανέκαθεν υπογράμμιζε την ανάγκη ε, απαλλαγή ε, των μεταφορών από τι ανθρακούχε εκπομπές, γιατί σίγουρα οι μεταφορές εκπέμπουν σημαντικές ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα και θα πρέπει να λάβουμε κάποιες προτάσεις και μέτρα για να μειώσουμε τι εκπομπέ άνθρακα. Γι' αυτό και λέμε για κινητικότητα με χαμηλέ εκπομπέ άνθρακα. Μα ενδιαφέρουν όλα αυτά και είμαστε πολύ σοβαροί στην προσπάθεια. Και επίση έχουμε την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών που δεν γίνεται μόνο σε περιφερειακό επίπεδο αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θα πρέπει να έχουμε στο πλευρό μα και του άλλου παγκόσμιου εταίρους Μα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνο μα. Γιατί ούτε η φύση έχουν, έχει σύνορα, ούτε οι ουρανοί έχουν σύνορα και στις συζητήσεις που είχαμε στην, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας αλλά και της Ναυσιπλοείας, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια σας παρουσίασα την έκβαση των συζητήσεων που είχαμε στην ΕΚΑΟ και πόσο σημαντικό είναι ε, που διευκολύναμε μια πρωτοφανή ε, διατομεακή συμφωνία για τον περιορισμό των εκπομπών στην αεροπορία. Και τώρα που ε, συνεχίζεται το έργο βλέπουμε ήδη τα πρώτα ενθαρρυντικά και θετικά αποτελέσματα από την ψηφοφορία του Συμβουλίου της ΕΚΑΟ τον Ιούνιο και θα συνεχιστούν ε, οι συζητήσεις και το φθινόπωρο. Αλλά πιστεύω ότι προχωρούμε προς ένα παγκόσμιο σύστημα που θα είναι πολύ φιλόδοξο για τον περιορισμό των εκπομπών στις αεροπορικές μεταφορές. Και θέλουμε όλο περισσότερες χώρες που να προσυπογράψουν Ήδη έχουμε 75 και μέλη νομίζω. θα μπορούσα να ψάξω τον αριθμό, αλλά δεν χρειάζεται, δεν είναι αυτό το σημαντικό. Πάντως πάντα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και θα πρέπει να δημιουργήσουμε ικανότητες και στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε και αυτές να συγκλίνουν. Και σίγουρα δεν έχουμε φτάσει στο αποτέλεσμα, αλλά είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέβαλε ε, πριν την ψηφοφορία του Ιουνίου στο Συμβούλιο της ΕΚΕΟ και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και το φθινόπωρο ώστε να συνάψουμε παγκόσμια συμφωνία για τις ανέρες μεταφορές για την πολιτική αεροπορία. Και τον Απρίλιο ε, και στην Επιτροπή Προστασίας του Αλάσιου Περιβάλλοντος καταφέραμε να προωθήσουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο για τον περιορισμό των μεταφορών και στην αυτιλία και χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό τώρα όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε και στην πράξη και να προσέξουμε και τις λεπτομέρειες για να δούμε πώς θα οδεύσουμε προς το 2050 ώστε να έχουμε τις μεγαλύτερες δυνατές μειώσεις εκπομπών όπως υποσχεθήκαμε. Και σίγουρα είχαμε και την ευλογία της δικής της Επιτροπής ε, στη προσπάθεια να συνάψουμε διεθνείς συμφωνίες και θα προωθήσουμε την ε, τέτοιε διεθνεί συμφωνίε, γιατί χρειαζόμαστε παγκόσμιε ε, συμφωνίε ε, για τα θέματα του περιβάλλοντο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κινητικότητα με χαμηλέ εκπομπέ άνθρακα και τι υποδομέ που χρειάζονται. Ναι, πιστεύω ότι εδώ χρειαζόμαστε σίγουρα πιο δαψιλά κονδύλια και πρόσφατα είχαμε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση υπό την δική σας αιγίδα για να προωθήσουμε την, τα εναλλακτικά καύσιμα και σίγουρα ε, θα πρέπει να έχουμε καλύτερες υποδομές και για τα ηλεκτρικά οχήματα και για τα υβριδικά και για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε επενδύσει. Από τη μία έχουμε την οδηγία για, για τα εναλλακτικά καύσιμα και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε εφαρμογή της. Οπότε να μπορέσουν και τα κρατημέλη να επενδύσουν σε σταθμούς ε, φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ή σε τερματικά υγροποιημένου ε, φυσικού αερίου. Και έπρεπε να δούμε τι άλλα εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας, τι μηχανισμούς. Επίσης αναφέρθηκε το Ταμείο για την Καθαρή Κινητικότητα και εκεί είχατε δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερως και προωθήσατε αυτή την πρόταση. Και όπως είπατε, στην τελευταία συζήτηση που είχατε στην Επιτροπή σας, όταν ε, εξετάσετε τροπολογίες της ε, ε, έκθεσης πρωτοβουλίας, ακόμη οι λεπτομέρειες έχουν κολλήσει στην Επιτροπή, στην Νομική Επιτροπή, αλλά πρέπει να προωθήσουμε αυτό το ταμείο στο μέλλον για να έχουμε πιο ταχεία πρόοδο στα θέματα της καθαρής κινητικότητας. Η κυρία Φώστερ, σας ευχαριστώ και για τα δικά σας σχόλια. Σας ευχαριστώ και για τη συνεργασία που είχαμε. Ξέρω ότι θα μείνετε αρκετό καιρό εδώ, αλλά όταν φύγετε θα μας λείψετε πραγματικά, γιατί όπως είπατε από την αρχή ε, στήριξετε πολλές προτάσεις, άλλες τις κατακρίνατε, αλλά ήσασταν πολύ επικοδομητικοί στη συζήτηση και η συνεισφορά σας ήταν ανάκαθα πολύ χρήσιμη. Και εσείς αναφερθήκατε στο συνδέοντα στην Ευρώπη και στην ανάγκη ύπαρξη ε, σημαντικών μηχανισμών για την πρόωθηση των υποδομών. Είμαστε ε, συνεργάτες λοιπόν και θα πρέπει να αντιληφθούμε και τις ε, προκλήσεις που έχουμε. Έχουμε το 100% των κονδυλίων να έχουν ήδη αναλυφθεί ως υποχρεώσεις μέχρι τις αρχές του έτους. Βλέπετε τι μεγάλη συνεργασία έχουμε και τι Επιτυχία στους ε, χρήστες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό 261 για την πολιτική αεροπορία, μας είπατε ότι είναι, ήταν πολλές οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε προκειμένου να προχωρήσουμε στον κανονισμό αυτό και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι ήταν πραγματικά ατυχές που για μία ολόκληρη πενταετία δεν καταφέραμε να σημειώσουμε καθόλου πρόοδο. Παρ' όλα αυτά δεν μέναμε με σταυρωμένα χέρια, σας διαβεβαιώ. Προωθούσαμε το ζήτημα και κάναμε διαβήματα προς όλες τις προεδρίες. Είχαμε όμως πρόβλημα τον ορισμό της επικράτειας και αυτό δυστυχώς επισκέσε όλες τις συζητήσεις για, για τα άλλα θέματα της ε, αεροπορίας. Είχαμε μια σημαντική συμφωνία με την Ουκρανία για την αεροπορία. Όλα αυτά τα θέματα μας παρεμπόδισαν στη συνολική πρόοδο, πάντως εμείς συνεχίσαμε να υποβάλλουμε νομοθετικές προτάσεις. Και προχωρήσαμε και σε άλλους τομείς και θα πρέπει να το διευκρινίσουμε από τη στιγμή που θα έχουμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε εδώ, σίγουρα θα την εκμεταλλευτούμε. Γιατί και οι ενδιαφερόμενοι έχουν πολλές προσδοκίες ε, να διευκρινιστούν τα πράγματα. Και καλώς που μας υπενθυμίσετε τις κατευθυντήρες γραμμές που βοήθησαν και ε, διευκρίνησαν τα πράγματα και έτσι μπόρεσαν και αρμόδιες αρχές εφαρμογής ε, να βελτιώσουν την εφαρμογή τους. Αλλά δεν έχουμε μερικές φορές εναρμονισμένη ερμηνεία για τα επιμέρους θέματα. Και υπάρχουν ε, πολλές υποχρεώσεις του 261 που δεν έχουν ακόμη τηρηθεί. Μερικές φορές είναι υπερβολικές όμως αυτές οι υποχρεώσεις. Επίσης αναφέρεται στο πλαίσιο αυτό το ATM, κάτι που είναι πολύ σοβαρό και ήταν πολύ σοβαρή κατάσταση και το καλοκαίρι. Και σίγουρα είναι παράδεκτες ε, αυτές οι απροσδόκητες απεργίες. Τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο τα λεπτά καθυστερήσεων στην Ευρώπη ήταν περισσότερα από ολόκληρο το χρόνο του 2017, μέσα σε τρεις μήνες. Και όλοι ε, κάνατε αεροπορικά ταξίδια και ίσως όλοι υποφέρατε από αυτές τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Και είχαμε 20% των πτήσεων στην Ευρώπη το καλοκαίρι που σημείωσαν καθυστερήσεις. Και αν δεν αλλάξει τίποτα θα έχουμε τα ίδια και του χρόνου. Αναφερθήκατε στις α, α, απροειδοποιητές απεργίες και όντως α, πολλές αεροπορικές εταιρείες μίλησαν για αυτό που επηρέασαν τις πτήσεις τους και οδήγησαν σε καθυστέρηση. Το καλοκαίρι μόνο οι απεργίες ήταν το 9% των αιτίων της, των καθυστερήσεων. 30% των καθυστερήσεων οφειλόταν στον καιρό και το υπόλοιπο 69% ήταν ικανότητες στο προσωπικό. Δύο στις τρεις σε δύο από ε, τους τρεις ε, κλάδους. Σε δύο από τους τρεις ε, τόπους κυρίως. Και για το σύνολο του 2017 οι ικανότητες της τελέχωση 56% μέχρι τον Αύγουστο ε, ε, και ο καιρό ήταν πολύ σημαντικότερο λόγο καθυστερήσεων από ότι οι απεργίε. Ο βασικό όμω λόγο, το βασικό έτοιμο των καθυστερήσεων ήταν οι ικανότητε στη στελέχωση. Δεν έγινε επαρκή προγραμματισμό για του ελεκτέ ενέργεια κυκλοφορία και για τι ε, υπηρεσίε ε, ε, στα αεροδρόμια. Αυτέ είναι οι βασικέ προκλήσει που θα αντιμετωπίσει και στο μέλλον η αεροπορία. Κύριε Τελίτσκα, παρακαλώ επισπεύστε κάπως γιατί Έχουμε, έχουμε και άλλο γύρο ερωτήσεων. Είχαμε μάλλον πολλές ερωτήσεις. Ε, κύριε Τελίσκα, ε, είχαμε σημαντική πρόοδο στον κανονισμό 868. Ξέχασε και το, τη μεγάλη συνεισφορά του κυρίου Πίπερ στο ζήτημα αυτό. Ελπίζω να το ολοκληρώσουμε μέχρι τα τέλη του έτους και για τον δίκτυ συνδεσιμότητας τον βελτιώνουμε και θα συνεχίσουμε να τον ενημερώνουμε. Ο κύριος Νταλούντε μίλησε για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και πώς θα δώσουμε ενάψματα στον κόσμο να χρησιμοποιεί το τρένο. Όντως για τις ε, μικρές αποστάσεις καλύτερα να χρησιμοποιεί το τρένο ο κόσμος. Αλλά όντως ε, ο κλάδο έχει βελτιωθεί γιατί για πολύ καιρό ήταν πολύ απρόθυμο στη χορήγηση των ε, στοιχείων. Κάτι που δυσκόλευε τον προγραμματισμό των ταξιδιών. Δεν είχαμε νέα συστήματα κρατήσεων εφάμιλα με αυτά τη αεροπορία. Αλλά και στις σιδηροδρόμου αλλάζουν τα πράγματα και χάρη σε εσά ε, σε μεγάλο βαθμό. Γιατί χάρη στο τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο ε, θα ρίνουμε τι εταιρείε να δίνουν τα στοιχεία τους και έχουμε και πιο εκλεπτισμένα συστήματα, πια πιο αξιζητημένα για τις μεταφορές. Και τώρα με τη, με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων μπορεί να γίνει και καλύτερος προγραμματισμός του ταξιδιού. Και είχαμε και πολλές προτάσεις που θα τις συνεχίσουμε και στο μέλλον, γιατί και εμάς μας ενδιαφέρει ε, η βελτίωση και η μεγαλύτερη χρήση των σιδηροδρομικών μεταφορών, γιατί ε, είναι και πιο προβλέψιμο και πιο αξιόπιστο το τρένο και πιο προσιτό στον κόσμο. Η κυρία Νταμάτο μίλησε για το συνδέοντα στην Ευρώπη και την Νότια Ευρώπη. Συμφωνώ απόλυτα ότι στη Νότια Ευρώπη θα θέλαμε περισσότερες επενδύσεις στις υποδομές του ΣΕΦ, του συνδέοντα στην Ευρώπη. Αλλά αυτό επαφίεται τη εθνικέ κυβερνήσει. Αυτέ αποφασίζουν πώ θα χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια του συνδέοντα στην Ευρώπη και των άλλων διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Δεν θα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κάθε κράτο που θα ε, χρησιμοποιήσει τα κονδύλια και τα TEN-T καλύπτει όλε τι χώρε και σχεδόν όλε τι περιφέρειε. Και από τη στιγμή που έχουμε κονδύλια στα δίκτυα TEN-T, στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, περιμένουμε τα κράτη-μέλη να υποβάλουν προτάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη και τη συνοχή και την ε, συνεκτικότητα στη συγκεκριμένη χώρα. Σε ό,τι αφορά τους ενιαίους εθέρες, ε, τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεις βάρος της ασφάλειας. Σίγουρα η ασφάλεια είναι η πιστή προτεραιότητά μας σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση, κανένα συμβιβασμό στην ασφάλεια. Και μάλιστα φέτος στην Ευρώπη ε, είχαμε 7,4 εκατομμύρια πτήσεις που απογειώθηκαν και προσγειώθηκαν με ασφάλεια. Και έχουμε υψηλά επίπεδα ασφάλειας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που δεν, ε, θα κάνουμε συμβιβασμούς. Και στο επόμενο πακέτο θα εξασφαλίσουμε τα υψηλά επίπεδα διαφάνειας. Ε, ασφάλεια, Με συγχωρείτε, αλλά έχουμε καθυστερήσει κιόλας. Δίνω το λόγο στην κυρία Μπάχ. Ένα λεπτό όμως μόνο. Καλώς ευχαριστώ κύριε Χαλολάη για τα όσα είπατε αλλά και για τους επένους στην Επιτροπή μας και την ε, σαφή τοποθέτηση ε, και επανατοποθέτηση των στοιχείων για τις απεργίες. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Ο κύριος ε, Ερτού, λοιπόν, ο συναδελφός, πολύ σωστά μίλησε νωρίτερα για τα κοινωνικά ζητήματα των απασχολουμένων στις αερομεταφορές, μίλησε για τις αυθαίρετες ή ε, επισφαλείς θέσεις εργασίας, για ντάμπινγκ, για μελέτες, πάνω απ' όλα. Και θυμάμαι και μια μεγάλη εκδήλωση με παρουσία και της Επιτρόπου Μπούρτς και της Επιτρόπου Τάισεν, που, για την οποία όμως λόγος δεν γίνεται. Συνέχεια δεν έχει δοθεί σε αυτά τις ε, μελέτες και τις ε, συζητήσεις. Θέλω λοιπόν να δω πιο συγκεκριμένες προτάσεις για τις αεροπορικές μεταφορές. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχω πολλά θέματα. Θα μιλήσω μάλλον πολύ γρήγορα προειδοποιώ. Ε, σε σχέση με την κοινωνική πτυχή της κινητικότητας, είναι ξεκάθαρο ότι έχει αποτύχει η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στο πρώτο στο πακέτο της κινητικότητας και καλό θα είναι να μην παρεμβαίνει στο κοινοβουλευτικό χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν το Κοινοβούλιο δεν ήταν σε θέση πριν το τέλος του χρόνου να υιοθετήσει θέση, τι θα κάνετε. Θα αποσύρετε τις προτάσεις σας και θα ξανακαταθέσετε μετά καινούργιες. Στην κινητικότητα επίσης έχουν αρχίσει οι υπηρεσίες σας να μελετούν μια νέα πρόταση για τον κανονισμό για τον χρόνο ανάπαυσης προλαμβάνοντας ενδεχομένως ε, αδυναμία λήψη απόφαση επίπεδο Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και τρίτον έχετε συνομιλήσει με κοινωνικού εταίρους για θέματα θεμελιώδη των συνδικαλιστικών σωματείων οργάνωση χρόνου εργασίας παραδείγματα. και γιατί όχι να γίνει και μια μεγάλη διαβούλευση με τους πολίτες για τα κοινωνικά ζητήματα των εργαζομένων στους, στο χώρο των μεταφορών. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο για όλους. Και επίσης η περιβαλλοντική πτυχή. Έχετε κάποιες προτάσεις ή σχόλια για, για τα σχέδια της, ευρωπαϊκής της Προεδρίας σε σχέση με τα διόδια, τα οδικά διόδια και για πότε το έχετε να καταλήξουμε συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ, Λοντότσκι. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Έχω ερωτήσεις για το πακέτο της κινητικότητας. Σε λίγο οι συντονιστέ μα θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουμε τι εργασίε για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία πάντως τον Ιούλιο έδειξε ότι ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά, ούτε οι συμβαστικέ τροπολογίε συγκέντρωσαν πλειοψηφία. Οπότε δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία να καταλήξουμε σε συμβαστικέ προτάσει για την απόσπαση εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση. Πριν από δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διέκοψε ε, τις ε, διαδικασίες επί παραβάση κατά της Γαλλίας και της Γερμανίας γιατί το Κοινοβούλιο επεξεργαζόταν ένα lex specialis σε μια ειδική νομοθεσία. Δεν νομίζω να προλάβουμε πάντως να το ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος της αιτίας οπότε θα επαναφέρεται εκείνη τη διαδικασία κατά των δύο χωρών, Γαλλίας και Γερμανίας. Νομίζω ότι Τήρησα το χρόνο μου, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρικέ, έχετε το λόγο ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και έχω δύο ερωτήσει: εκ των οποίων η πρώτη είναι σχετικά με το Brexit, ε, γεγονός στο οποίο δεν χρειάζεται να επανέλθω. Ε, ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν διαφόροι διορθωτικοί κανονισμοί στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, μπορεί το Κοινοβούλιο να μην συμμετέχει ευθέω στη συζητήση, αλλά θα έχει τη τελική και καθοριστική ψήφο για την τελική ε, πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να επιτρέψει και πώς την Επιτροπή Μεταφορών να συμμετάσχει στην ε, συζήτηση για τα θέματα των μεταφόρων και πώς, ε, ανεξάρτητος μάλιστα του υλικού αποτελέσματος, πώς ε, πιστεύετε ότι μπορείτε να το εξασφαλίσετε αυτό. Επίσης μιλήσατε για το MIE, για τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, ποια εικόνα έχετε σε σχέση με τα θέματα των μεταφορών και τη δυνατότητα, κομμάτι της ανταγωνιστικότητας να πάει στο MIE, δηλαδή όχι κινητικότητα, αλλά μια οργάνωση. Ο κύριος Κράμερ. 10 στόχοι, 14 πρωτοβουλίες είχαμε ακούσει πριν από μερικά χρόνια. Τι συνέβη εν τέλει. Επίσης, ανώτερα βία στα δικαιώματα των ε, καταναλωτών ή επιβατών. Η Ryanair πολύ συχνά ε, επικαλείται την ανωτέρα βία και λέει ότι δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει, να αποζημιώσει. Ωστόσο ευτυχώ το γερμανικό ανώτατο δικαστήριο κατέριψε αυτά τα επιχειρήματα και την υποχρεώνει σε αποζημίωση. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να διαδοθεί γενικώ και όλοι να συμπεριφέρονται όπως οφείλουν. Επίσης, ε, μια και έχουμε να κάνουμε χρήματα, η ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία της επέκτασης των σιδηροδρομικών δικτύων στην Ευρώπη, θα πείσετε τις ε, χώρες να κλείσουν μικρά κενά που υπάρχουν και που δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση των δικτύων. Στη Γερμανία από το Κότμπους ε, μέχρι τα προνοϊκά σύνορα 150 ε, χιλιόμετρα έχουν μείνει ανολοκλήρωτα και πρέπει να κλείσουν. Το ίδιο Βρυξέλλες Βαλονσιέν. 800 μέτρα είναι το κενό που μας λείπει για να ολοκληρωθεί το δίκτυο και να περιορίσουμε από τις δύο στη μία ώρα τη διάρκεια της διαδρομής. Πώς θα πιέσετε, πώς θα εξα... Ε, τα κράτη αυτά να κάνουν τη δουλειά τους. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Δελή. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και σύντομες ε, παρατηρήσεις, συμφωνώ απολύτως και με εσάς κύριε Χολολάη και με τους συναδέλφους εδώ ότι η Τετάρτη Ιουλίου δεν ήταν και τόσο μνημειώδης εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είχαμε πολλά να χαιρετήσουμε. Ωστόσο ρωτώ, τι βλέπετε ως δυνατότητα κινητικότητας. Εγώ ήμουνα ε, εισηγητή στο τέταρτο πακέτο για του σιδηροδρόμους και δεν θα ήθελα να ξαναδώ σενάριο αντίστοιχο με αυτό που αντιμετωπίσαμε στην τέταρτη δέσμη για του σιδηροδρόμου. Θα θυμάστε φαντάζομαι ότι είχαμε ετοιμάσει, είχε ετοιμάσει η προηγούμενη θητεία, η προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. ε, μια πρώτη ανάγνωση, μετά άλλαξαν πολλά στις θέσεις του Συμβουλίου, ήρθε να αλλάξει το κείμενο του Κοινοβουλίου, πολιτικές αντιπαραθέσεις δεν έγιναν όπως έπρεπε και ήταν μεγάλη αποτυχία. Βλέπετε λοιπόν κάποια κινητικότητα σε επίπεδο Συμβουλίου. Και μια άλλη ερώτηση για τη διαδική χρήση των δικτύων TNT. Ε, δεν βλέπετε κάποια δυνατότητα να αντιμετωπιστούν ή κάποια πιθανότητα να εμφανιστούν προβλήματα χρηματοδότησης και πώς μπορούμε αυτά να τα προβλέψουμε, τι είδους κατευθύνσεις μπορούν να πάρουν και πού μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Ευχαριστώ. Βλέπετε κάποια απειλή δηλαδή από εκεί. Ευχαριστώ κυρία Γκραπίνη για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και κύριε Χολουλάη, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την παρουσίαση Βλέπουμε ότι γεμίζει σιγά σιγά το ποτήρι σε σχέση με την, με την συνδεσιμότητα. Ε, λέτε ότι τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση της, ε, να προβούν στις επιλογές για τις υποδομές. Αλλά έχω να ρωτήσω το εξή εάν χορηγούνται από, την Ευρωπαϊκή, από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό κονδύλια στα κράτη-μέλη Πώς μπορούμε να μην απαιτούμε να λειτουργούν οι υποδομές στα ανατολικά κράτη-μέλη κατά τρόπο ισοδύναμο με αυτά των δυτικών, των παλαιότερων κρατών μελών, γιατί υπάρχουν περιοχές ολόκληρες που δεν έχουν καν σιδηροδρομική γραμμή και έτσι δεν λειτουργεί ολόκληρο το δίκτυο. Μεταφορές. Εάν μεταφορές από μια δυτική προς ανατολική χώρα περνάμε μέσα από τρία διαφορετικά κράτη. Ε, ε, χρησιμοποιεί μεθόδους dumping με βάση χαμηλούς μισθούς, δεν πρέπει να το αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο. Ο κύριος Καπούτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να ε, βρίσκεται αντιμέτωπη για άλλη μια φορά με κινήσεις οι οποίες θα μπορούσαν στον τομέα των μεταφορών ακόμα και να αναιρέσουν τη μείωση του, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Πρέπει να βρούμε λοιπόν νέες προδιαγραφές σε σχέση με τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται. Πρέπει το κοινό κέντρο έρευνας ε, να δώσει ε, στοιχεία για το ότι ορισμένοι παραγωγοί προσπαθούν να ε, παρουσιάσουν τεχνητά στοιχεία για τις εκπομπές των καυσαερίων φουσκώνοντα τα τωρινά στοιχεία εκπομπών και ω εκ τούτου εξουδετερώνοντα η αδίποτε πρόβλεψη για μείωση εκπομπών στο, στο μέλλον με αυτά τα τεχνητά στοιχεία. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τον ε, Γενικό Διευθυντή τη ε, Γενική Διεύθυνση MOVE ε, και εν ώψη των χαμηλών εκπομπών ε, άνθρακα, τι σκοπεύει να κάνει απέναντι σε αυτό την ε, προσπάθεια που για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε να παρουσιαστούν ψευδή στοιχεία από την αυτοκινητοβιομηχανία. Ευχαριστώ, Ντεμόντε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω βέβαια με τα όσα είπε και η Επίτροπο, η Πρόεδρος νωρίτερα για το ΙΓΕΦΕΡΑ της Γένοβα θεωρώ πολύ λυπηρό, για να μην πω αχαρακτήριστα τα όσα λυπηρά και αχαρακτήριστα τόσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης όπου σε ένα δυστύχημα που χάθηκαν 43 ανθρώπινες ζωές βρήκε τρόπο να αξιοποιήσει για λόγους εσωτερικής προπαγάνδας εις βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης την τραγωδία και θα ήθελα να ρωτήσω συγκεκριμένα τι είδους δυνατότητες βλέπετε ε, έργο σε παραχώρηση αυτοκινητοδρόμου να ε, προχωρήσει στην αποκατάσταση και επισκευή με πρώτο μέλημα βέβαια πάντα την, την ασφάλεια. Αυτό. Ε, επίσης ε, αερομεταφορές Ryanair έχει προσελκύσει τους, τους προβολείς της δημοσιότητας λόγω των απεργιών, ωστόσο βλέπουμε ότι βρίσκει τρόπους να αρνηθεί την ε, αποζημίωση των επιβατών. Πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατέψει τα δικαιώματα των επιβατών. Η Πρόεδρος ευχαριστώ. Κύριε Αντεμόντε, κύριε Ολολάη, έχετε πολύ λίγη ώρα για να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Όχι, γιατί δεν έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε Ολολάη, όπως πριν. Έχετε όμως αρκετά ερωτήματα να απαντήσετε. Πολύ γρήγορα, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. και ευχαριστώ πολύ τις κυρίες και κυρίους βουλευτές για τις ερωτήσεις. Ενδεχομένως να μην εξαντλήσω τις απαντήσεις, ίσως και γραπτός θα πρέπει να συμπληρώσω κάποια ζητήματα, εάν θεωρήσετε ότι δεν είναι επαρκείως λεπτομερείς οι απαντήσεις μου. Για τον κύριο Μπάχα, και ζητώ συγγνώμη που χρειάστηκε να επαναλάβετε μια ερώτηση που είχε που είχε ήδη διατυπωθεί αλλά την ώρα που ετοιμαζόμουν να δώσω αυτή την απάντηση, διαπίστωσα ότι είχε λήξει ο χρόνο μου και αναγκάστηκα να σταματήσω. Ναι, βεβαίω, βεβαίω είναι πάρα πολύ σημαντική η κοινωνική διάσταση, οι κοινωνικέ διατάξει στι εναέρειε μεταφορέ. Είναι πολύ σημαντική και η στρατηγική μα και άρα πρέπει να κάνουμε κάτι έτσι ώστε όλα τα κοινωνικά δικαιώματα ε, των οποίων χαίρουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να επεκτείνονται και στις εναέριες μεταφορές, όπως συμβαίνει άλλωστε γενικά. Έχουμε μια αιτήση Έχουμε μια μηνιαία συνάντηση διμερή ε, όπου συζητούμε όλα τα κοινωνικά ζητήματα με τους εμπλεκόμενους φορείς και βεβαίως ε, τα κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν. Ε, έχουμε άλλωστε αναθέσει και μελέτη, την αναφέρατε κι εσείς, όπου ζητούσαμε προτάσεις για συγκεκριμένα βήματα ή συγκεκριμένες αλλαγές στους, στην ισχύουσα νομοθεσία το 2008 ε, και πάνω απ' όλα εντοπισμός της έδρας του home base. Ε, άπαξ και καθοριστεί αυτό, νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε πολλά άλλα συναφή ζητήματα. Μια έκθεση θα δημοσιευθεί στο τέλος του χρόνου με πολλά θέματα ε, και βέβαια της, ε, την απασχόληση, αλλά αυτό μέχρι ότου ολοκληρωθεί η μελέτη που έχουμε αναθέσει ε, δεν μπορούμε να το κάνουμε παρά μόνο να διαπιστώνουμε ότι 18% ε, των πιλότων και 20% του λοιπού πληρώματος ε, απαντά σε ερωτηματολόγια μας ότι προσλαμβάνεται πλέον με ατυπικές μορφές απασχόλησης και πρέπει να δούμε τι είδους γραμμή θα βρούμε για να καλύψουμε όπως πρέπει τις ανάγκες αυτές. Ε, άλλωστε και ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το επισημάνατε όμω και εσεί, έχει πει ότι δεν πρόκειται να γίνει νέα νομοθετική πρόταση από την Επιτροπή μέχρι το τέλο τη θητεία. Επομένω, έκθεση πρωτοβουλία μην περιμένετε. Ωστόσο, διεξοδικότατη ανάλυση θα γίνει και θα είμαστε σε θέση είτε στο τέλος του έτους είτε στις αρχές του προσεχούς να υποβάλουμε τον προβληματισμό, την ανάλυση και αντίστοιχα και ένα ξεκάθαρο σχέδιο δράσης που θα προτείνει νέα βήματα από εκεί και πέρα. Αυτό για να σας δείξω με πόση σοβαρότητα βλέπουμε τα θέματα. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι σε πολλές περιπτώσεις ε, την ε, υλοποίηση την έχουν στα χέρια τους οι εθνικές αρχές. Και προσπαθούμε και εκεί που κάποια ζητήματα ίσως ε, είναι πιο ψηλά στην προτεραιότητα ορισμένων κρατών να βοηθούμε, αλλά και σε εκείνα που λιγότερο έχουν προτεραιότητα. Ο χρόνος βέβαια μας πιέζει πολύ. Κινητικότητα με πολλά ερωτηματικά και η κυρία Τεβός είπε ότι έχουμε, ότι πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις. Το θέμα όμως δεν είναι οι πιέσεις. Είναι βέβαιο ότι όλοι θέλουμε να βρούμε λύση. Και θα την ε, περιέγραφα την πίεση αυτή ως θετική πίεση, γιατί συμφωνούμε όλοι πως η κατάσταση όπως έχει τώρα είναι χειρότερη από αυτό ε, που θα μας εξασφάλιζαν οι συμβασμοί. για το πρώτο πακέτο που έχουν συμφωνηθεί. Και όπως είπα, ε, είμαστε στη διάθεσή σας ε, επί 24 ώρου βάσεως. Εάν υπάρξει ανάγκη, αν υπάρχει ανάγκη για υποστήριξη. Το ζήτημα είναι αν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε απόφαση μέχρι το τέλος του χρόνου. Και αν δεν τα καταφέρουμε, αποσύρουμε, αποσύρουμε την πρόταση. Όχι, εάν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν αποσύρουμε την πρόταση. Αυστριακή Προεδρία. και πρόοδος στα περιβαλλοντικά στοιχεία. Ναι, βεβαίως, βεβαίως και συνεργαζόμαστε με την Προεδρία της Αυστρίας και βεβαίως προσπαθούμε και σε αυτούς να ασκήσουμε αυτή τη θετική πίεση. Προσβλέπουμε σε πρόοδο. Όμως είναι περιορισμένος και ο χρόνος μας και το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Οπωσδήποτε σε αυτούς τους τομείς στους οποίους θα είναι δυνατόν να ληφθούν ε, αποφάσεις, να γίνουν επιλογές και ξέρουμε ότι και εμείς θα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Η Αυστριακή Προεδρία αυτή τη στιγμή έχει αναπτύξει διμερείς επαφές, λεβόμενη το ε, θερινό διάλειμμα ε, μπαίνουμε και εμείς στο παιχνίδι και περιμένουμε μέχρι το τέλος του μήνα συμβαστικές προτάσεις από την Προεδρία στο Συμβούλιο για να διαμορφωθεί μια εικόνα σχετική με το Συμβούλιο όπου ξέρουμε ότι τα πράγματα έχουν τις ίδιες δυσκολίες να αντιμετωπίσουν όσο και εδώ. Όμως και δυνατότητες βλέπουμε για επίτευξη λύσης. Και πιστεύω ότι πρέπει κανείς να εγκαταλείψει τις ακραίες θέσεις ε, από κάθε πλευρά γιατί είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται, όχι ακραίε επιθυμίε, αλλά ακραίε ω προ τα προτινόμενα. Γιατί δεν πρόκειται ούτε η μία ούτε η άλλοι ε, άκρα να κερδίσουν. Και άρα θα πρέπει να περάσουμε σε μια πιο κεντρική ε, λύση που θα έχει πιθανότητες να καταλήξει σε συγκεκριμένη πρόταση. Υπάρχουν ζητήματα τόσο αλληλέντατα που δεν μπορεί κανείς να απομονώσει στο ένα και να πει προχωρώ στη λύση αυτού αλλά εγκαταλείπω το άλλο. Όλα αυτά λοιπόν συνενωμένα συγκερασμένα μπορούν να δώσουν ένα καλό αποτέλεσμα. Πιστεύω, Χωρί βέβαια να θεωρώ ότι θα είναι κάτι εύκολο αυτό. Ο κύριος Λοτόφσκι επίση μας ρώτησε για, τις για την ενεξελίξη διαδικασία παραβάση. Βεβαίως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, είναι ε, επιτάπητος οι προτάσεις μας, δεν έχουμε τίποτε αποσύρει, παραμένουμε ε, παραμένουμε στις θέσεις μας, παραμένουμε δηλαδή στην επεξεργασία του, προγρά... του πακέτου για την κινητικότητα. Δεν νομίζω όμως ότι εάν δοθεί λύση πρέπει απαραίτητα να συνεχίσουμε με σκληρό τρόπο να ε, ε, συνεχίσουμε τη διαδικασία παραβάση. Αλλά εάν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακας των συνθήκων θα πρέπει να ε, κάνει το καθήκον της και να συνεχίσει τη δικασία επί παραβάση. Για τον κύριο Ρικέ και το Brexit έχουμε δύο προτάσεις ε, για την προπαρασκευή που ανέφερα και νωρίτερα. Στη συναπόφαση ε, θα έρθουν, οπότε εσείς θα συμμετάσχετε ως Επιτροπή πλήρως στην επεξεργασία των προτάσεων. Βεβαίως ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος με όλα τα θέματα που έχουμε εκκρεμεί, δημοσιονομικοί περιορισμοί, και δυνατότητες για επενδύσεις στις ε, υποδομές. Βεβαίω το συνδέοντας στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό, αλλά έχουμε και τα περιφερειακά ταμεία, το κοινωνικό ταμείο, πολλές δυνατότητες για επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αξιοποιήσει ο τομέα των μεταφορών. Ένα 12% νομίζω των έργων συνολικά μπαίνουν μέσα στο χώρο των μεταφορών, αλλά υπάρχουν διάφοροι τρόποι να συνδυαστούν τα ποσά το πολύ καλό ε, του συνδέοντας στην Ευρώπη είναι ότι χορηγεί χρηματοδότηση ε, με, με δωρεά και όχι μορφή δανείου και έτσι ε, μπορεί να εξασφαλίσει την ανέγερση υποδομών και εδώ τα ποσά αυτά πρέπει να διατίθενται προκειμένου ακριβώς να κλείσουν τα κενά, δηλαδή να συνδεθούν τα δίκτυα ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν τα κομματάκια τα μικρά στους σιδηροδρόμους ή να ανοίξουν οι στενοποί. Πολύ σωστά λέει ο κύριος Κράμερ ότι υπάρχουν τμήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα οποία δεν έχουν γίνει επενδύσεις και ξέρω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο επανελειμμένως επαναφέρεται χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Κράμερ. Ναι, βεβαίως το έχουμε επισημάνει και εμείς στις συνομιλίες μας με τα κράτη-μέλη αλλά τελικά είναι η επιλογή των κρατών μελών, των ίδιων. Όμως τους λέμε, να, έχετε το συνδέοντα στην Ευρώπη, έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε αυτό το κενό στο δίκτυο, γιατί να μην το κάνετε. αυτό ανεξαρτό του συγκεκριμένου παραδείγματος που αναφέρατε εσείς, μην ε, ε παρανοηθώ παρακαλώ. Θα πω όμως ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν κλείνει το κενό αυτό στο δίκτυο για να μην επιτραπεί η ανάπτυξη ενός ανταγωνισμού που κάποιος δεν θα ήθελε να βρει μπροστά του. Δεν είναι δηλαδή αδιανόητο αυτό, αδιανόητος αυτός ο σχεδιασμός. Ξέρουμε ότι σε μεγάλο βαθμό εγκαταλείφθηκε ο σειροδρόμος για να μην επιτραπεί να μπει κάποιο άλλος στην αγορά. Λευκή βίβλος, θα πρέπει να επανέλθω. Ε, με λεπτομέρειες γιατί δεν έχω ακριβή στοιχεία για το πόσα έχουμε επιτύχει και πόσα όχι. Πριν από τέσσερα χρόνια είχαμε μια αξιολόγηση που πιστεύω αποδεικνύει πως είναι ακόμα χρήσιμη η Λευκή Βίβλος. Έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Τώρα δεν ξέρω αν λέω πιο πολλά από ό,τι πρέπει, αλλά θεωρώ ότι έχει έρθει πια η ώρα η προσεχής επιτροπή να ε, μελετήσει την ε, ε, επεξεργασία μιας νέας λευκής βίβλου. Όπως είπα, έχει κάνει πολλά, ε, μπορεί να αποτελέσει ένα, ένα πλαίσιο για να χτίσουμε ε, στους διάφορους τομείς των μεταφορών επιπλέον, αλλά όπως είπα δεν θέλω να ξεπεράσω τα εσκεμένα. Έχετε ξεπεράσει κατά τρεις φορές το χρόνο που σα είχα δώσει, τα τρία λεπτά που σα είχα δώσει, έχουμε φτάσει στα 10 λεπτά και 30 δεύτερα, αλλά επειδή ακολουθεί μια συνεδρία των συντονιστών, υποχρεούμε να σας διακόψω. Ε, τι λοιπέ απαντήσει θα δοθούν γραπτό. Σας ευχαριστώ θερμά για την ε, ε παθιασμένη απάντηση σε ερωτήσεις. Ας ε, χειροκροτήσουμε τον κύριο Ρολάι.